Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίζουμε τώρα. Ε, θέλετε να κάνουμε έναν έλεγχο πρώτα απ' όλα για να δούμε την παρουσία σας. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για να τσεκάρουμε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, υπέρ κατά αποχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι η Ενωτική Αριστερά θα καταθέσει έκθεση μειοψηφία, λέει ο κ. Κόσο Περμούη. Μάλιστα, ναι, το έχουμε σημειώσει αυτό, το έχουμε υπόψη μα. Αρχίζουμε. Έχουμε τον κατάλογο ψηφοφορία. Είστε όλοι παρόντες. Ωραία, τροπολογία παριθμών 1 έχει αποσυρθεί. 30 και 38 ψηφίζουμε μαζί, υπέρ, κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Επανάληψης. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Όχι ακόμα, περιμένουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ποιος δεν ψηφίζει. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 96. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 100. Ψήφι Κατά. Παρακαλώ να χέρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116 και 117 μαζί είπε. κατά αποχές εγκρίνονται. 118. Α, όχι, όχι, αποσυρθεί. 119 και 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 Υπε Α, όχι, καταπίπτει. Συμβαστική 3 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 122 είπε. κατά Αποχές. Θεωρώ ότι έχει εγκριθεί. 124 είπε, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 Είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 Check. Ωραία. Επαληθεύουμε την τροπολογία 141 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Όλα εντάξει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 153. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και θα περάσουμε τώρα σε τέσσερις ταυτόσημες 158 μέχρι 161 υπέρ, κατά, αποχές, δεν σηκώνεται χέρια. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 165 γιατί οι υπόλοιπε καταπίπτουν. 165 είπε. Κατά. άποχε. Εγώ θα έλεγα ότι έχει απορριφθεί μάλλον. Τσεκ, καλά. Θα την ελέγξουμε λοιπόν. 165. Πέρας. Δεν κρίνεται. Παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας λίγο πιο ψηλά. 166, 67, 168, 169, 170, 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 172 όχι έχουν καταπέσει αυτές 175-176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 177 υπέρ κατά αποχές Αυτό χρειάζεται έλεγχο, παρακαλώ. 177. Αρχίζει ψηφοφορία και τελειώνει κιόλας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ σηκώνετε λίγο πιο ψηλά τα χέρια σας, σας βλέπω. 179 υπέρ. Συγγνώμη, 178 λέει ο πρόεδρος υπέρ. Όχι, έχει καταπέσει. Με μπερδεύει εδώ η γραμματεία. 179. Καταπίπτει τώρα ή δεν καταπίπτει. This one doesn't fall if the is before the adopted. This is reference to this. Okay, third one. Okay. No, it falls. 179. 179 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τι έγινε με την 178. Ρωτάει κάποιος. Όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε την 178. Λοιπόν, υπέρ της 178. Τροπολογία 178. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα, συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές 220 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 221 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 222 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. 222. And vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 225 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαλήθευση για τη 225. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 239 υπέρ, καταπίπτει, συγγνώμη. Όχι, δεν καταπέπτει. Check on 238. Λήθευση για τη 238. Άρχεται η ψηφοφορία. We close the vote. Πέρας. I'm a bit too quick. We close the vote. ψηφοφορίας. Εγώ δεν ψήφισα, αλλά ούτω ή άλλω απορρίπτεται. 239 υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 241 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 243 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Για την 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23-24 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά.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 Αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση. Vote is open. Vote is closed. ψηφοφορίας εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Ξανά υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 79 περ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81, 82, 83, 84, 85 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 αποσύρεται, 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Αποσύρεται. Συγγνώμη, δεν ψηφίζουμε, είναι γλωσσική. 3 υπέρ, κατά, ξανά, υπέρ, Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Για την τρία, πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Υπέρ και πάλι για τέσσερα, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα να κάνουμε μια επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, βλέπω την ίδια πλειοψηφία, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαλήθευση για την 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάλι με την ίδια πλειοψηφία. Υπέρ. Όχι για την 8. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε τώρα το σύνορο του κειμένου ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is Εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, στην εισηγήτρια. Περνάμε τώρα στο σημείο 11. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία με αυτό. Να ευχαριστήσω του συναδέλφου και αν σκοπεύετε να αποχωρήσετε, ησύχω παρακαλώ. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 11 στην ημερήσια διάταξη. Πρώτη συζήτηση της γνωμοδότησης για την αναδιατύπωση του κανονισμού για τα είδη διπλής χρήσης. Η αρμόδια επιτροπή επιτροπή είναι ίντα και η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι η κυρία Μαριώτη Χάκε. Προθεσμία, παρακαλώ ησυχία. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών σε δύο μέρες, 4 ε, Μαΐου στις 2 η ώρα. Θα δώσω το λόγο στην, στην της χρωμοδότησης για την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε λίγο ησυχία, αλλιώς θα χρειαστούμε λίγο χρόνο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και λίγο τεχνικό το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν την υπομονή σας. Χαίρομαι που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτή τη γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής ΑΦΕΣ για τα αναδιατύπωση κανονισμού ειδών διπλής χρήσης που συζητούμε στην Επιτροπή ΙΝΤΑ. Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στην ε, πρώτη γραμμή, είτε πρόκειται για την ασφάλεια, είτε για τεχνολογικά στοιχεία. Πρέπει να δώσουμε δυνατότητες ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μετριάσουμε και τις απειλές. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωση ω ε, υπεύθυνο και παγκόσμιο παράγοντα για την διάδοση τεχνολογιών που δεν αφορούν μόνο τα ε, συμφέροντά μας αλλά και τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα παγκοσμίω. Είναι πολύ σημαντική η επικαιροποίηση, διότι έχουμε πολύ γρήγορε τεχνολογικέ εξελίξει και αλλάζει συνεχώ η παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή προσέγγισε το θέμα από την οπτική γωνία της ασφάλειας των ανθρώπων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγγνώμη, συνάδελφοι, κύριε Καστάλτο, σας παρακαλώ. Είναι πολύ δύσκολο, με συγχωρείτε η αναδιατύπωση και επικαιροποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν, διότι έχουμε πολύ γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές και αλλάζει και η ισορροπία των δυνάμεων σε γεωπολιτικό επίπεδο. Υποστηρίζω με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να βάλουμε στο επίκεντρο την ασφάλεια των ανθρώπων, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, για την αναδιατύπωση αυτή. Θεωρώ επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις σε τομείς ε, στους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φρόντισε να είναι αρκετά σαφή πρέπει να ευθυγραμμίσουμε περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις εξωτερικές και στις εμπορικές πολιτικές και να φροντίσουμε να υπάρχει συνοχή με των πολιτικών και των μέσων ασφαλείας που διαθέτουμε και να υπάρχει και ισορροπία σε σχέση με τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντά μας. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε και κάποιες τεχνολογίες ε, παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, ε, ήδη διπλής χρήσης, ε, διότι αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για διάπραξη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για τα συμφέροντα που έχουμε σε θέματα ασφαλείας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν χρειάζεται έλεγχο κάθε νέα τεχνολογία και η εξαγωγή τεχνολογιών που μπορούν να ενισχύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία τους, όπως για παράδειγμα η κρυπτογράφηση, θα πρέπει να ενισχυθούν και όχι να τα ελέγχουμε χωρίς λόγο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει περιττό άχθος για τους εξαγωγείς και να υπάρχουν περαιτέρω γραφειοκρατικά προσκόμματα όταν πρόκειται για έρευνα στο διαδίκτυο, για παράδειγμα. Ο στόχος λοιπόν της ασφάλειας και το, η τελική χρήση κάποιων αγαθών είναι πάρα πολύ σημαντικός για να μην έχουμε παράνομες μεταφορές από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ασφάλεια δικαίου. Ε, κυρίως ε, η τεχνολογία παρακολούθησης στο κυβερνοχώρο χρησιμοποιείται και για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και για να διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο κάποια σοβαρά δικήματα στη συνέχεια ε, για παράδειγμα παράνομη απόκτηση πληροφοριών ανθρώπων που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή δημοσιογράφους όταν παίρνουμε στοιχεία από τον υπολογιστή τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία στρέφονται κατά των μελών της αντιπολίτευσης για την κράτησή τους, φυλάκησή τους κλπ. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όχι μόνο το γεγονός ότι αλλάζει η πραγματικότητα επιτόπου για κάποιες χώρες, αλλά και υπάρχουν και επαναστατικές τεχνολογικές αλλαγές ε, γύρω μας, ε, τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη. Όταν λοιπόν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ε, συγκεκριμένα προϊόντα διπλής χρήσης, θα πρέπει να είναι ελεγχόμενες αυτές οι διαδικασίες και θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε διαδικασίες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις αλλαγές επιτόπου σε τρίτες χώρες ή στις τεχνολογικές αλλαγέ. Ολοκληρώνω λέγοντα ότι ε, οι ξένες συναλλαγές γίνονται όλο ένα και πιο περίπλοκες, επομένω πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών και να ενισχύσουμε και τη διαφάνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις πληροφορίες της αδειοδότησης για να υπάρχει κατάλληλος έλεγχος και υποπτία. και επίσης ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, διότι κάποιοι ακόμα το κάνουν σε θελοντικό επίπεδο. Ε, για την παραβίαση του κανονισμού θα πρέπει επίσης να είναι πιο ομοιόμορφες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναδιατύπωση αυτή ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό ε, από την Αραβική Άνοιξη και τις εξεγέρσεις εκεί. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό το τεχνολογικό ζήτημα και να συνεργαστούμε επικοδομητικά ώστε να είναι πολύ σημαντικό και για τώρα αλλά και για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Ο κύριος Ντανζόν για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να προσθέσω πολλά σε αυτά τα οποία μόλις είπαν ε, η, η, είπε η συγγήτρια. Είναι σαφές ότι η πρότασή της ακολουθεί την σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο Ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να δούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δεν θα πρέπει εμείς μονομερός να τους προσθέσουμε βάρη τα οποία δεν αναλαμβάνονται από ανταγωνιστές τους σε άλλες χώρες ε, φιλελεύθερες και δημοκρατικές. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αθέμητος ανταγωνισμός και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένα σαφές ε, πλαίσιο νομικό, ιδιαίτερα για το άρθρο 4 που προτείνει ε, την διεύρυνση του πεδίου της ρήτρα catch all. Ε, πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε λίγο τα πράγματα διότι σε επίπεδο τρομοκρατίας αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ότι στην συγκεκριμένη έννοια της τρομοκρατικής δράσης ε, να γίνονται αυτές οι δράσεις με, ε, με βασικές πρωτόγονες μορφές τεχνολογίας. Τα προϊόντα διπλής χρήσης λοιπόν που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι πραγματικά ατελείωτο, δηλαδή όπλα αλλά και αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συγκεκριμένοι και να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το άρθρο 4. Υπάρχουν επίσης κάποιες άλλες διατυπώσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο ενίσχυσης και διευκρίνησης ε, ε, για την ορολογία τους εννοώ, όταν όμως μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή θέση. Ευχαριστώ κύριος Μάρτιν για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ την Μαρίτσα για τη δουλειά της. Από τη μία δεν είναι εύκολο να μπορέσει κανείς να ορίσει την δυτή χρήση στον τομέα ας πούμε της τεχνολογίας ελέγχου και τεχνολογίας παρακολούθησης. Από την άλλη όμως, κάνοντας το αυτό δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις και εδώ οι κυβερνήσεις πρέπει να προσέξουν και να μην απαιτήσουμε από τις μικρομεσαίες να αναλάβουν υπέρογκα βάρη. Θα πρέπει λοιπόν και να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σεβαστούμε τα οικονομικά μας συμφέροντα. Εμείς νομίζουμε ότι ο όρος και ο ορισμός που χρησιμοποιούνται για τις τεχνολογίες παρακολούθησης δεν είναι ο σωστός. Επίσης η διαδικασία παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι συγκεκριμένη δεν διευκρινίζεται το τι είναι η σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με την απλή σε εισαγωγικά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, σχετικά με την δέουσα επιμέλεια, προφανώς θα πρέπει και αυτό να το ορίσουμε κάπως καλύτερα. Οι ορισμοί αυτοί είναι θεμελιώδεις για τις επιχειρήσεις που απαιτούν για να λειτουργήσουν μια κάποια νομική σταθερότητα. Συνεπώς λοιπόν εμείς λέμε ότι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρότασή μας είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά απαιτούνται περισσότερες διευκρινήσεις πριν γίνουν δεκτές οι προτάσεις της. Τώρα για το να μην επιβαρύνουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι σαφές αυτό. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση όμως να είμαστε συνένοχοι εξαγωγής προϊόντων διτής χρήσης που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να πιέσουμε τις άλλες χώρες να σεβαστούν τα δικά μας επίπεδα προστασίας και όχι εμείς τα δικά τους. Για τους πράσινους τώρα. Η κυρία Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Μπούχνερ είναι ο σκιώδης εισηγητής μας ε, των Πρασίνων και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2010 συστηματικά ζητούμε να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την εξαγωγή αγαθών διτής χρήσης. Γιατί είχαμε και πολλά σκάνδαλα. Λοιπόν, παγίως εμείς ζητούσαμε επιτέλους ε, όταν εξάγουμε ε, υλικό παρακολούθησης και τεχνολογίες να ε, το ελέγχουμε. Είναι ψηφιακά όπλα αυτά που μπορούν να προκαλέσουν τεράστια απειλή και είναι και και ζημία μάλλον και είναι και απειλή για τις ανοιχτές κοινωνίες. Δεκαπέντε ε, φορές πιέσαμε ε, μόλις πέρσι. Τώρα έχουμε την ευκαιρία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε το καθεστώς εξαγωγών και πώς θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Μπορούμε να δείξουμε τώρα ότι 15 ψηφίσματα της Ολομέλειας που απαιτούσαν κάτι τέτοιο γίνονται πραγματικότητα και με τη δυνατότητα να αλλάξουμε και την πραγματικότητα. Υποστηρίζουμε λοιπόν καταρχήν ε, την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα για το σχέδιο ε, της κυρίας Χάκε και εδώ υποστηρίζουμε τις προτάσεις σας και μάλιστα στεναρά και πλήρως. Και βεβαίως η γνωμοδότηση αυτή θα έρθει να βελτιώσει και να ενισχύσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για μας είναι καθήκον της Επιτροπής ΑΦΕΤ να έχουμε μια εξωτερική πολιτική ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο και θα κάνουμε προτάσεις ακριβώς για να ενισχυθεί αυτή η διάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών. Η συγγήτρια θέλει να επανέλθει για κάποια συμπεράσματα. Θέλω. Πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Χονδρικά είμαστε στην ίδια γραμμή όλοι. Με τις δικές μου τροπολογίες, τι προσπαθώ να κάνω, ακριβώ να διευκρινίσω τους ορισμούς. Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά, όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τους διάφορους οργανισμούς, ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι θεσμοί έχουν κάποια κριτήρια και κάποιους ορισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, αυτά ήδη έχουν θεσπιστεί. Ή όταν πρόκειται για την τρομοκρατία, που είναι πολύ ευρία έννοια και πολύ εύκολο να πέσει σε καταχρήσεις, υπάρχει κοινή θέση του Συμβουλίου, στην οποία παραπέμπουμε και αναφερόμαστε, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και γιατί κυρίως δεν μιλάμε. Ε, υπάρχει κανένα κενό που άφησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι τα εργαλεία της παρακολούθησης ε, στον κύβερνο χώρο και αν αυτό ε, χρησιμοποιείται με την ένεση του χρήστη ή χωρίς αυτή. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν υπάρχει Κάποιο που κάνει μια έρευνα και θέλει να έχει πρόσβαση στο κινητό μου για να το κάνει πιο ασφαλές, δίνω τη συνένεσή μου. Εάν όμως ερήμην μου και εναγνία μου κάποιο παίρνει στοιχεία από το κινητό μου και τα χρησιμοποιεί αργότερα, δεν παραβιάζει μόνο το δικαίωμα στην ιδιωτική μου ζωή, αλλά ε, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο για να παραβιάσει και άλλα δικαιώματά μου. Θα βρούμε τρόπους πρακτικούς για τους ορισμούς, για να μην είναι πολύ ευρύς και γενικοί, για να αποφύγουμε διπλωματικές ευαισθησίες, που είναι και αυτό ε, ε, μέλημα της δικής μας Επιτροπής, και να μην επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους. Συμφωνώ με τον David Μάρτιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει ηγετική στάση εδώ, να βάλει ψηλά τον πύχη και να πείσει και άλλες χώρες να την ακολουθήσουν, γιατί αυτό είναι σοβαρό θέμα ε, της διάδοσης αυτών των υλικών δεν είναι μόνο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα αλλάζει το τεχνολογικό τοπίο. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις ε, και ενωτόμου τρόπους καταστολής διαπιστώνουμε δυστυχώς σε άλλα μέρη του κόσμου. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Όπως σας είπα προηγουμένως, ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι στις 5 Μαΐου, λέει ο Πρόεδρος, στις 12 το μεσημέρι και στις 29 το μηνός θα το ξανασυζητήσουμε ενώ ε, θα εγκριθεί στις 30 Μαΐου για να πάει στην Επιτροπή Ίντα και στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Ολοκληρώνεται εδώ το σημείο 11 στην ημερήσια διάταξη και προχωρούμε στο 12 πολιτικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία. Ένα σχέδιο έκθεσης Είναι πολύ σημαντική η Ινδία και η στρατηγική μας ε, σχέση αυτό φάνηκε από αποστολή της Επιτροπής μας το Φεβρουάριο. Είπε ότι εκπρόσωπο Μογκερίνη πριν από δύο εβδομάδες μετέβη στη χώρα επίσης εν ώψη ε, της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας που θα διεξαχθεί στο Νέο Δελχή. Η έκθεσή μας θα εγκριθεί στην Ολομέλεια πριν το θέρος. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πρέντα, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι. Χίλια ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας ε, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι μακρά ιστορία, πολύ πλούσια, πολύ σύνθετη επίσης. Έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά επίθετα για να συνοψίσουν αυτές τις σχέσεις. Έχουμε πει ότι κάποιοι λένε ότι είναι φυσική σχέση, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι στρατηγική σημασία, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι απόλυτα εδρεωμένες αυτές τις σχέσεις ε, και ε, υπάρχουν και κάποιες αναφορές οι οποίες λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία έχουν μια σχέση η οποία θεμελιώνεται βάσει αξιών. Αυτό είναι ο κατάλογος λοιπόν των χαρακτηρισμών που χρησιμοποιούνται. Η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας είναι ε, όλα αυτά μαζί και θα έλεγα ότι κυρίως πρόκειται για μία σχέση που έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες και πολύ σημαντικές προοπτικές για το μέλλον. Οι προκλήσεις ε, ε, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ινδία είναι παρόμοιες ε, τη σήμερον ημέρα και στον οικονομικό τομέα. Υπάρχουν περιφερειακές εντάσεις αλλά και ε, παγκόσμιας προβλήματα όπως η τρομοκρατία, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και φυσικά η κλιματική αλλαγή. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι η αυξημένη συνεργασία και συντονισμένη δράση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας ε, μόνο θετική μπορεί να είναι και για τις δύο πλευρές. Ε, θεωρώ ότι θα ήταν ιδανικό η, συνεργασία αυτή να πάει πέραν της οικονομικής συνεργασίας και βεβαίως οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Ε, ο στόχος της έκθεσής μου σήμερα είναι να εκφράσουμε την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια πιο στενή εταιρική σχέση και πιο ισχυρή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας. Βεβαίως αυτή η εταιρική σχέση θα πρέπει να ενισχυθεί σε πάρα πολλούς τομείς, στον οικονομικό τομέα, ε, στον περιβαλλοντικό τομέα, αλλά ε, στον πολιτιστικό τομέα. Κυρίως ενδιαφερόμαστε στην έκθεση για την ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία λόγω της φύσης της, έκθεση, Επιτροπής μας. Υπάρχει και η αποστολή την οποία μόλις αναφέρατε, ε, το ταξίδι που έκαναν κάποια μέλη της Επιτροπής μας ε, το Φεβρουάριο στο Νέο Και από την έκθεσή μου θα ήθελα να εκφράσω τρία μηνύματα τα οποία ελπίζω να είναι σαφή. Το πρώτο ε, είναι ότι όσον αφορά εμάς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή για την έγκριση μιας στρατηγικής για τη σχέση μας με την Ινδία γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε μια συνεκτική πολιτική. Και πάλι από πλευρά μας θα πρέπει τους επόμενους μήνες και χρόνια να φροντίσουμε να υπάρχει καλύτερο συντονισμός μεταξύ κρατών μελών και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής για να επιτευχθούν οι στόχοι μα ε, με καλύτερο τρόπο και πιο εύκολο τρόπο και βεβαίως αυτό το οποίο αντιλήφθηκα και επιτόπου είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ινδία. Ε, δεύτερο μήνυμα θα ήθελα να ε, χαιρετήσω την ε, τρίτη διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας το 2016 και ε, κάποιους φιλόδοξους στόχους για τη συνεργασία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί αυτό το θεματολόγιο και μάλιστα αυτό ανέφερε και η κυρία Φεντερίκα Μογερίνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθορίσουμε συγκεκριμένα βήματα και να δοθούν συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. Όπως είπατε και εσείς, η κυρία Μογερίνη μετέβει προσφάτως στην Ινδία και είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό για να αναπτύξουμε και τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας να γίνονται ε, τακτικά αυτές οι σύνοδοι κορυφής. Ε, προτείνω λοιπόν να γίνει και το φθινόπωρο και να αυξηθούν οι σύνοδοι κορυφής για να υπάρχουν ανταλλαγές ε, σε υψηλό επίπεδο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Όταν συναντηθήκαμε με τους εταίρους μας της Επιτροπής Εξωτερικών Θεμάτων του Ινδικού Κοινοβουλίου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και από πλευρά του ενδιαφέρον να γίνονται πιο τακτικές επαφές και να υπάρχει και κατάλληλο συντονισμό σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Τρίτο μήνυμα για τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. Θέλησα να επισημάνω κάποιους ε, άξονες εργασίας, τους οποίους θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία δεν έχουν πάντα την ίδια θέση, αλλά ε, ο ειλικρινής και τακτικός διάλογος μπορεί να είναι υποφελής και για τους δυο μας και να μπορέσουμε να επιτύχουμε και τους κοινού μας στόχους. Είτε πρόκειται για το Αφγανιστάν, είτε για την Κίνα, είτε τη Ρωσία, ε, σίγουρα μπορούμε να συνεισφέρουμε με συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε ουσιαστικά τις εντάσεις σε θέματα ασφαλείας και στην Ασία αλλά και στα περίχωρα της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικός λοιπόν αυτός ο άξονας, θα πρέπει να υπάρχει πιο στενή συνεργασία και ε, στην παράταση της δήλωσης που έγινε για το θέμα αυτό στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Θεωρώ επίσης ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία είναι αναφανδόν υπέρ ε, μιας ε, διεθνούς πολυμερής συμφωνίας, ε, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε από κοινού τις θέσεις μας στα διεθνή βήματα για να τονίσουμε αυτές τις κοινέ μας προοπτικές και προσδοκίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι επειδή υπάρχουν κοινέ αξίες θα πρέπει να προβάλλουμε περαιτέρω το ρόλο αυτό στην εταιρική σχέση που θέλουμε να έχουμε. Υπότιτλοι Authorwave ε, οι σχέσεις αυτές βέβαια δεν εξαντλούνται στους άξονες που σας ανέφερα και ούτε και η έκθεση είναι πλήρης βεβαίως επειδή δεν υπάρχει περισσότερος χώρος. Το γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει αυτός ο προεριορισμός. Προτείνω λοιπόν μέσω τροπολογιών να περιλάβουμε και άλλους τομείς όπως για παράδειγμα ανταλλαγές ε, σε επίπεδο σπουδαστών ε, στην επιστημονική έρευνα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθεί η έκθεση στην Ολομέλεια εγκαίρως, δηλαδή τον Ιούλιο, ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνδίας, η οποία προβλέπεται για το φθινόπωρο. Ελπίζω λοιπόν οι τροπολογίες σας να είναι επικοδομητικές και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στενά με τους κοιόδης συζητητές προκειμένου να μπορέσουμε μέσω από αυτή την έκθεση να ε, δώσουμε μια ισχυρή όθηση στις κοινέ μας σχέσεις με την Ινδία. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στους κοιόδης συζητητές. Η κυρία Γκίλη είναι στον κατάλογο μόνο από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες από ό,τι βλέπω και από πλευρά σκιωδών να τη δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Κριστιά για μια πολύ ισορροπημένη πρόταση. Όπως είπες Κριστιά, Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες διαθέσιμες για την ολοκλήρωση της έκθεσης αυτής και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν και πάρα πολλές δυσκολίες. Πάντως οι σχέσεις έχουν αρχίσει να βελτιώνονται με, την, με την κυρία Μογκερίνη και μάλιστα στη συνάντηση που είχαμε στο Δελχή πριν δύο εβδομάδε, πράγματι συμφώνησε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο συχνά σε πάρα πολλού τομεί όπως η άμυνα, η θαλάσσια ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική δράση κτλ. κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλό αυτό να ακολουθηθεί με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και έχω την αίσθηση ότι θα συμφωνήσω μαζί σας όταν πείτε ότι η ετήσια συνάντηση κοροφής την οποία είχαν στο παρελθόν θα συνεχιστεί έτσι ώστε στο Δελχή πάλι τον Ιούνιο να δούμε ακριβώς οι τομείς αυτοί σε ποιο βαθμό έχουν σημειώσει πρόοδο βλέποντας το τι συμβαίνει παγκοσμίω, αυτός ο διάλογος είναι ιδιαίτερος επίκαιρος. Όταν συνδυάσει κανείς τα θέματα αυτά με την πολιτική ε, των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των διεθνών οικονομικών σχέσεων, καθίσταται σαφές ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε χρόνο και θα πρέπει να επενδύσουμε πολιτικά για να καλύψουμε τα κοινά του παρελθόντος. Η συμφωνία αυτή, η εταιρική, είναι μια καλή πρόταση. Θυμίζω ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ινδία ξεκίνησαν εδώ και 10 χρόνια. Από το 2013 όμως μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Μια χώρα η οποία κατέχει στρατηγικό χώρο σε μία περιοχή η οποία θα εκπροσωπεί το 60% της ε, μέσης τάξης στον κόσμο μετά το 2020. Τον Φεβρουάριο που είχαμε πάει στην Ινδία ε, δείξαμε ότι σαν κοινοβούλιο αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει, ιδιαίτερα βλέποντας τι γίνεται και με τους δύο Ινδούς εργαζόμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα προς το παρόν και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει δυνατότητα όλων μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας με την Κίνα, υπάρχουν ε, ε, σχέσεις και εντάσεις οι οποίες σε αυτή τη φάση δεν βρίσκονται στο καλύτερο θα έλεγα σημείο. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να δούμε και τι εταιρικέ συμφωνίες μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων και της ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να επιταχύνουμε τον διάλογό μας και να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις. Το Δελχή έχει διεκδικήσει μία μόνιμη θέση στο Συμβουλίο Ασφαλείας, θυμίζω. Η συνεργασία με την Ινδία επίσης στην Αφρική, στον Ινδικό, θα πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερα στον τομέα καταπολέμησης της πειρατείας. Υπάρχουν και άλλα θέματα, τα οποία τέθηκαν όταν πήγαμε εκεί όπως ε, η αντιμετώπιση της βίας ε, ε, στα πλαίσια της έμφυλης αντίληψης, όπως επίσης και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΛΟΑΤ, έχει σημασία να έχουμε μια αντιμετώπιση η οποία να επιδιώκει αποτελέσματα συγκεκριμένα και μόνο μέσω της επίτευξης των αποτελεσμάτων αυτών θα βελτιώσουμε τον διάλογο γενικότερα σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι η έκθεσή σας λοιπόν θα βοηθήσει στην ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης η οποία θα προωθήσει ακόμα περισσότερο τα κοινοτικά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ και σκοπεύω να συνεχίσουμε την συνεργασία μας και στις τροπολογίες και στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι σκιώδεις παρόντες σε αυτή τη φάση. Περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών. Θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά σε αυτούς που το ζήτησαν. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριος Πέτερλε, δεν θα έλεγα ότι ανήκω στους ε, φωτεινούς ε, ομιλητές αφού εξαντλήσαμε τους σκιώδεις. Ε, όλοι φωτεινοί και λαμπροί είμαστε όταν συζητούμε για τις σχέσεις μας με την Ινδία. Ευχαριστώ την εισηγητή τον κύριο Πρέντα που ε, δεν ακρηγόρησε αλλά έτσι με φιδό χρησιμοποίησε τις βασικές έννοιες από την αρχή και μιλάει για ε, πιο ισχυρές και πιο βαθιές σχέσεις με την Ινδία. Συμφωνώ απολύτως. Εγώ ξέρετε ότι είμαι εισηγητής για την στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. Και όπως γνωρίζετε, διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, εμπορική και ελευθέρου εμπορίου, αλλά και στρατηγική ε, συμφωνία και εταιρική σχέση και μέχρι στιγμής είναι 40 οι τομείς στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε περιγράψει στις ε, διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Και εκτός αυτών, 8 ε, ειδικοί τομείς έχουν εντοπιστεί, ειδικά θέματα όπου επιθυμούμε να συνεργαστούμε. Εκτός των 40 δηλαδή. Συμφωνώ ε, και με τα όσα είπε η κυρία Νίνα Γκίλ. Θέλουμε περισσότερο δυναμισμό στις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και περισσότερη φιλοδοξία, γιατί εκεί χωλένουμε, θα πρόσθετα εγώ. Και οι πρόσφατες εξελίξεις μας δίνουν νέα επιχειρήματα, θα έλεγα, για περισσότερη δυναμική και πιο δυναμική προσέγγιση. Και αν δεν γίνουν αυτά πριν την επόμενη Σύνοδο Κορυφή, ελπίζω στην Σύνοδο Κορυφή αυτή να δοθεί η απαραίτητη όθηση ε, σε αυτή τη συνεργασία και να πυροδοτηθεί αυτή η προσπάθεια, να επιταχύνουμε και με μεγαλύτερη φιλοδοξία. Ένα τελευταίο. Μεταξύ των 40 τομέων στρατηγικής συνεργασίας με την Ιαπωνία, Έχουμε εντάξει και την υγεία. Για πρώτη φορά νομίζω εντάσσεται σε μια στρατηγική συμφωνία ο τομέας της, υγείας. Και για ποιο λόγο να μην έχουμε και με την Ινδία τέτοια ε, στρατηγική συνεργασία, όχι μόνο λόγω Αγιουρβέντα, που είναι γενικά παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η Ινδική Ιατρική, αλλά θέλουμε μια δυναμική και φιλόδοξη προσέγγιση και υποστηρίζω την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπασίρ από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας, κύριο Πρέντα, για την εξαιρετική του έκθεση, που είναι ισόρροπη, θετική και βρήθη συγκεκριμένων ε, συστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία όντως θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους προς το συμφέρον της ευημερία και της ασφάλειας ε, που θα σφυριλατήσουν στις περιφέρειές τους η καθεμιά αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Για να ενισχυθεί λοιπόν μια έκθεση που είναι ήδη πολύ καλή και μελετημένη, θα ήθελα να προσθέσω εγώ να προτείνω τα εξή σημεία. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι η Ινδία έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, με στόχο αυτή η αχανής χώρα να γίνει παλόμενη δημοκρατία ε, χωρίς αποκλεισμούς η κοινωνία. Αυτό είναι ένας ευγενής στόχος και μεγάλη πρόκληση. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά λέγει η έκθεση, παραμένουν βάσιμες ανησυχίες ε, λόγω των διακρίσεων με βάση την κάστα, αλλά και την μη βέλτιστη μεταχείριση απέναντι σε μειονότητες και εθνικές και θρησκευτικές ομάδες. Εγώ είμαι αναφαδόν υπέρ του ελευθέρου εμπορίου και της ελεύθερης αγοράς. Ε, υποστηρίζω πλήρως ε, όλες τις πτυχές για μια ευρύτατη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Ωστόσο, ε, το ελεύθερο εμπόριο και ελεύθερη αγορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό στο τελικό κείμενο. Το Πακιστάν έχει πληρώσει βαρύ τίμημα υποστηρίζοντας τη Διεθνή ε, Συμμαχία κατά των Ταλιμπάν και της τρομοκρατίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ινδίας και όλων των γειτονικών να ενισχύσουν το συντονισμό τους ε, σε όλη την περιοχή της Νότιας Ασίας. Ερχόμενος τώρα στις διμερείς σχέσεις Ινδίας-Πακιστάν. Το παρόν κείμενο και πάλι είναι πάρα πολύ εύγλωτο και πάρα πολύ εύσχημο, αλλά θα πρέπει να τονίζουμε ιδιαίτερα το εξής. Δεν χρειάζεται προσέγγιση μόνο για να είναι βιώσιμη η ειρήνη μεταξύ των δύο μεγάλων αυτών εθνών. Η ειρήνη δεν είναι αυτός σκοπός από μόνη της. Χρειαζόμαστε την ειρήνη έτσι ώστε να οικοδομήσουμε ε, ανάπτυξη, βιώσιμη και ευημερία που να φτάνει μέχρι και το τελευταίο πρόσωπο και το τελευταίο άνθρωπο σε αυτή την περιοχή. Και εδώ συμπεριλαμβάνεται και το Κασμίρ που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα Το Κασμίρ που βρίσκεται υπό την ειδική διοίκηση υπολείπεται κατά πολύ ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανάπτυξη σε σχέση με το Κασμίρ του Πακιστάν. Ας είμαστε λοιπόν ε, θαραλέοι και πούμε ότι όσο χειραφετούνται οι αυτόχθονες πληθυσμοί για να ευημερούν τόσο το καλύτερο για όλους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα είχαμε δώσει και το λόγο στην Υπηρεσία εξωτερική δράση, αλλά δεν φαίνεται ότι έχουμε κάποιον εκπρόσωπο εδώ για να μιλήσει εκ μέρου του. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πρέντα, αν θέλει να σχολιάσει. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητά το λόγο. Κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ ούτε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ούτε η... κάποιος εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ινδίας. Ε, δεν ξέρω, μπορεί να γιορτάζουν ακόμα την Πρωτομαγιά, κρατάει λίγο παραπάντα. κρίμα, αλλά γιατί είναι, είναι σημαντικό το ζήτημα για όλες τις πολιτικές ομάδες. Τώρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Είμαι αισιόδοξο διότι διαπιστώνω ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις, όχι μόνο από πλευρά σοσιαλιστών, που εξακολουθούν να είναι τμήμα αυτού του μεγάλου συνασπισμού που διαπραγματευτήκαμε στην αρχή της αιτίας, αλλά και ο σκιώδης ε, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών μου έστειλε ένα μήνυμα και τον ευχαριστώ για τα λόγια του και ο κύριος Βανόρντεν, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα, μου έστειλε ένα μήνυμα για τη σημασία της συνεργασίας για να μπορέσουμε να έχουμε συνένεση επί του θέματος αυτού εν αναμονή των τροπολογιών αν συμφωνήσει και ο πρόεδρος ο Ντέβιτ Μακάλιστερ να μπορέσουμε να ψηφίσουμε λίγο νωρίτερα θα ήταν πάρα πολύ καλό. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το οργανώσουμε βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ όλους και ελπίζω να μην βρεθώ με 900 τροπολογίες. Δηλαδή όσοι θέλουν να προσθέσουν κάτι το οποίο έχουμε βάλει σε χίλιες άλλες εκθέσεις να μην ε, κάνουμε τέτοια πράγματα. Καλό είναι να περιοριστούμε στις πολιτικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας και όχι τα χιλιάδες θέματα που συζητάμε ως Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ε, φταίει ο τρόπος που διεξάγονται τη συζήτηση, αλλά όλοι θέλουν να προχωρήσουμε. Θα το θεωρήσω ως ε, τιμή. Φάνηκε ότι την τελευταία φορά είχαμε δυσκολίες γιατί είχαμε πολλές εκθέσεις, ε, τίθεται και θέματα καθυστέρησης μετάφρασης. Η υπηρεσία μας θα δει τι δυνατότητες υπάρχουν. Δεν ε, φαίνεται όμως και πολύ ε, εύκολο. Είμαστε όμως πολύ αποτελεσματικοί σήμερα και εν γέννη ως Επιτροπή. Να ευχαριστήσω λοιπόν όσους έλαβαν το λόγο και να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 5 Μαΐου, 12 η ώρα και το χρονοδιάγραμμα είναι το γνωστό προς το παρόν. 19 Ιουνίου η ε, δεύτερη συζήτηση θα ψηφίσουμε στις 20 Ιουνίου και στην ε, Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία. Με αυτό ολοκληρώνουμε και το σημείο 12 και πάμε στο σημείο 13. Ενημέρωση για την ε, αποστολή στην Παλαιστίνη, ε, της αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη. Είχαμε επίσκεψη στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ στις 20 με 24 Φεβρουαρίου. Η αντιπροσωπεία ζήτησε, αλλά δεν έλαβε άδεια για να επισκεφθεί τη λωρίδα της Γάζας. Κανονικά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιτρέπεται να επισκεφθεί τη λωρίδα της Γάζας και επομένως περιμένουμε και κάποια νεότερα γι' αυτό να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για την ε, σχέση με την Παλαιστίνη για να μας ενημερώσει για την ε, αποστολή και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Αντιπροσωπείας. Ε, κύριε Σιλικιώτη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώσουμε για την αποστολή στην Παλαιστίνη. Ε, πριν να προχωρήσω στην Παλαιστίνη για την ε, αποστολή, θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας στην απεργία μπίνας που ξεκίνησε στις 17 Διδάκτου από 1.500 φυλακισμένους Παλαιστίνους στις φυλακές του Ισραήλ. Η απεργία συνεχίζεται μέχρι αυτή τη στιγμή και οι φυλακισμένοι Παλαιστίνοι ζητούν διασφάλιση βασικών δικαιωμάτων τους όπως αυτό της επίσκεψης της οικογένειας και τον τερματισμό της κράτησης τους χωρίς κατηγορίες ή δίκη. Θα ήθελα η Επιτροπή αυτή να συνταχθεί με την αντιπροσωπεία μας και να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων. Σα καλούμε επίση να σταλεί κατεπηγόντω η ερευνητική αποστολή για άμεση εκτίμηση τη κατάσταση στο φυλακισμένο. Όσον αφορά την αποστολή, η αποστολή τη αντιπροσωπείας έλαβε χώρα τον περασμένο Φλεβάρι. Συναντήσαμε τον Πρωθυπουργό Χαπτάλα και άλλου υπουργού. Είδαμε επίση ομόλογου μα από το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο. Είδαμε επικισμούς να οικοδομούνται, επιπλέον τη γη η οποία σηματοδοτείται και προρίζεται για μελλοντική επέκταση των επικισμών. Πισκεφτήκαμε αγροτικές κοινότητες των οποίων τα σπίτια και τα σχολεία βρίσκονται υπό απειλή κατεδαφίσεων. Εν ολίγης, είδαμε την υφέρπουσα αποσάρτηση της δυτικής όχθης να επιτυχάνεται καθώς η κατοχή εισέρχεται στο 50ο έτος της. Συγκλονιστική στιγμή κατά την αποστολή μα αποτέλεσε η επισκεψή μα στο στρατιωτικό δικαστήριο του Όφερ, όπου είδαμε να δικάζονται παιδιά ηλικία ακόμη και 13 ετών. Εκεί βιώσαμε μια πραγματική τραγωδία. Είναι συγκλονιστικό το πώ μπορεί ένα παιδί να βιώνει την κατάσταση αυτή. Η αντιπροσωπεία μα δεν θα πάψει να αγωνίζεται για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και των βασικών ανθρώπινων ελευθεριών κάθε παιδιού. Ακόμη είδαμε ένα ευρύ φάσμα συνομιλητών από διάφορες γενιές, κοινότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίοι μας μετάφεραν την αυξημένη τους απογοήτευση στο καθεστώς φιλετικού διαχωρισμού, το οποίο βιώνουν καθημερινά, αλλά και στην απουσία της προοπτικής στη λύση δύο κρατών. Η στήριξη στη λύση δύο κρατών είναι ακόμη κυρίαρχη, αλλά κάποιοι εκ των συνομιλητών μα διατύπωσαν τη σκέψη και στη λύση ενό κράτου. Ακόμα και ο Πρωθυπουργό Χαπτάλα είπε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να σκεφτεί τη λύση ενό κράτου εάν εγκυάται αυτή η λύση ίσα δικαιώματα για όλου του Παλαιστινίου. Για την ακρίβεια, οι φωνέ που μίλησε για τη λύση ενό κράτου αποτέλεσαν και ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα τη αποστολή μα. Ακόμα ένα αξιοσημείωτο εύρημα ήταν το εξή. Τεχνικά, η συγκρότηση του Παλαιστινιακού κράτου έχει ολοκληρωθεί χωρίς όμως να είναι πραγματικό κράτος. Η Παλαιστίνη υπό αυτές τις συνθήκε δεν μπορεί να κάνει καμιά πρόοδο και τα θεσμικά όργανα του κράτους θα κατεκαιρματιστούν και η κατάσταση θα χειροτερέψει όσο δεν προχωρούμε στη λύση δύο κρατών. Το ευρωπαϊκό έργο επιτόπου στην Παλαιστίνη, το οποίο είδαμε κάποια πολύ καλά παραδείγματα που αφορούν την ανθρωπιστική πλευρά, δεν στοχεύει ε, τελικά στην ουσιαστική πρόθεση της ευρωπαϊκής πολιτικής υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό εναπόκειται κυρίως στο Συμβούλιο και ότι η Επιτροπή παλεύει με τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά χρειάζεται να τονίσουμε πως χωρίς ουσιαστική πολιτική βούληση για την πρόθεση της λύσης δύο κρατών η ευρωπαϊκή πολιτική επιτόπου δεν θα καταφέρει πολύ περισσότερο. Οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να δείχνουν εκπληκτική αντίσταση σε όλη τη σκληρότητα τη καθημερινότητά του. Το γεγονό αυτό δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να διαγράψει όλε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν καθημερινά, αλλά και ούτε από τον πραγματικό κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται η λύση των δύο κρατών. Από του συνεχόμενου αυξανόμενου επικισμού, αλλά και από την έλλειψη ελπίδα και την απουσία τη ειρηνευτική διαδικασία. Συνεπώς ε, εμείς προτείνουμε τα εξής. Το πρώτο, μια πολιτική λύση είναι κατεπίγουσα. Επιβάλλεται πολιτική θέληση για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών πριν η ελπίδα χαθεί για πάντα. Καλούμε το Συμβούλιο να αποκτήσει ισχυρή θέση και να δράσει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή. Δεύτερο, η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν μπορούμε να ζητούμε λύση των δύο κρατών εάν δεν έχουμε δύο κράτη. Είναι γι' αυτό που καλούμε του συναδέλφους να εργαστούν άμεσα στα κράτη-μέλη του με τα κράτη-μέλη του για την αναγνώριση τη Παλαιστίνη. Τρίτον, η Παλαιστινιακή συμφιλίωση, η συγκρότηση κυβέρνηση τη Εθνική Ενότητα και οι εκλογέ είναι επιτακτική ανάγκη. Ένα δημοκρατικό κράτο δικαίου πρέπει να προχωρήσει στη διεξαγωγή αμερόληπτων εκλογών για όλα τα θεσμικά όργανα. Όσον αφορά την Παλαιστινιακή Αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει προσεκτική ώστε να διασφαλιστεί η καλή διακυβέρνηση, η διαφάνεια και ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαμορφώσει του όρου για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνέ δίκαιο σε οποιαδήποτε βοήθεια δίνει ή σε όποια εμπορική σχέση έχει στην περιοχή. Πέμπτον, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία των ΗΠΑ 2334 αποτελεί ξεκάθαρη έκφραση της διεθνούς πολιτικής συνένεσης ενάντια στους επικισμούς. Είναι μια βάση πάνω στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα πρέπει να δράσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τις πολιτικές πάνω στις νόμιμες της θέσεις, δηλαδή εδάφη πέραν της πράσινης γραμμής είναι κατεχόμενα πελαιστινιακά εδάφη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρεί σε οποιαδήποτε συμφωνία ή κοινά προγράμματα με το Ισραήλ σε γίνει η οποία εκτείνεται πέραν της πράσινης γραμμής. Οποιασδήποτε συμφωνίες με το Ισραήλ, περιβαλλοντωμένων και αυτών που είναι υποκύρωση, πρέπει να εγωδόνται τα σύνορα του 1967 και να περιλαμβάνουν ξεκάθαρες και ορθές εδαφικές ρήτρε. Οι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να παρακολουθούν στενά το ζήτημα αυτό. Το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη συνεχτική εφαρμογή των συμπεράσματων του Συμβουλίου Ασφαλείας και να αντιμετωπίσουν τυχόν κενά μεταξύ αυτών και τη πολιτική εφαρμογή. Οι κατευθυντήριε γραμμέ αναφορικά με τη σήμαση είναι ένα παράδειγμα αυτού του κενού. Η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει περισσότερε τι διάφορε και ω θεματοφύλαξη των συνθηκών να διασφαλίσει ότι ο νόμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται. Χρειάζεται ισχυρή και συλλογική δράση ενάντια στι κατεδαφίσει. Οι ανθρωπιστικέ προσπάθειε δεν αρκούσαν από μόνε του, Μόνο μαζί με την πολιτική δράση θα πετύχει ώστε η Παλαιστίνη να γίνει κράτος και να έχουμε τη λύση δύο κρατών. Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, τότε ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος για μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση. Πάνω σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε τα εξή. Την αύξηση του πληθυσμού και τον περιορισμό σε πηγές περιλαμβανομένης της γης, του νερού και της ενέργειας, στην, ε, ε, μέσω της κατοχής της Δυτικής Όχθης και του αποκλεισμού της Γάζας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε αυξημένες πιθανότητες ριζοσπαστικοποίησης, μετανάστευσης και βίας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την Ευρώπη, την περιοχή, καθώς και το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Και τέλος, ε, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει μαζί με τα κράτη-μέλη της και τους θεσμούς να δράσουν ώστε να καταστεί η λύση των δύο κρατών ζήτημα προτεραιότητας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση αυτή σχετικά με την αντιπροσωπεία στην Παλαιστίνη. Δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Για να το λέξω και πάλι. Όχι. Οπότε... σημειώνουμε τα όσα είπατε, θα εγγραφούν στα πρακτικά και σας ευχαριστώ πολύ που μας ενημερώσατε σήμερα. Ολοκληρώνεται το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης και προχωρούμε στο 14. Θέλει λίγη προετοιμασία. Έχουν έρθει οι ομιλητές μας. Έρχονται. Ωραία. Δύο λεπτά διάλειμμα για να περάσουμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα. <clears throat> now in Λοιπόν, βελτιωνόμεθα τεχνολογικά όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε το σημείο 14 τώρα μπροστά μας, το τελευταίο. Καταπολέμηση της ασυλίας, της ατιμορρησίας, ο ρόλος του διεθνούς ποινικού και τροπολογίες Καμπάλα στο καθεστώς της Ρώμης, στον κανονισμό συγγνώμη της Ρώμης. 5 Οκτωβρίου του 2016 αποφασίστηκαν. Το Διεθνές Ποινικό δημιουργήθηκε από την Συμφωνία της Ρώμης, η οποία τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιουλίου του 2002. διευρύνεται ή μάλλον διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής και η δικαιοδοσία του δικαστηρίου αυτού και ο ρόλος του σε περιπτώσεις επιθέσεων και εγκλημάτων πολέμου. Αλλά δεν είχαν ξεκαθαριστεί τα θέματα των επιθέσεων από χώρα σε χώρα και γι' αυτό στην Καμπάλα υπήρξε μια τροπολογία, η λεγόμενη τροπολογία Καμπάλα. Καθορίζεται το έγκλημα λοιπόν της επιθέσεως. Assembly Regulation 3314. E According to this amendment, acts of aggression ε, τέτοιου είδους δράσεις είναι η εισβολή σε άλλο κράτος, ο αποκλεισμός των λιμένων και των ακτογραμμών του, η επίθεση ε, σε επίπεδο υπηρετικής χώρας ή σε επίπεδο θαλασσίων ε, ε, περιοχών, η χρησιμοποίηση άτακτων ή μισθοφόρων εναντίον τρίτων χωρών και χρήση εδαφών από τρίτες χώρες που επιτίθενται σε μία πρώτη χώρα. Λοιπόν, η τροπολογία αυτή θα τεθεί σε λειτουργία ένα χρόνο μετά από την επικύρωση και λέγεται εδώ ότι εγκλήματα επίθεσης τα οποία διαπράττονται ένα χρόνο μετά από την επικύρωση ανήκουν πλέον στη δικαιοδοσία, δηλαδή 1η Ιανουαρίου του 2017. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και για την τροπολογία των 134 εμπλεκομένων χωρών, συμμετεχουσών χωρών μάλλον, οι οποίες θα αποφασίσουν να ασκήσουν την συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Έχουμε τρεις εκλεκτούς ομιλητές σήμερα για την πιθανή υιοθέτηση της τροπολογίας της Καμπάλα, η οποία θα επηρεάσει νομίζω εν πολύ στις εργασίες του δικαστηρίου. Η κυρία Πρόστ είναι υπεύθυνη του γραφείου του Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχει διάφορες υψηλού τύπου νομικές θέσεις. Ήταν ομπουτσμαν επίσης του Γενικού Γραμματέα ε, της Επιτροπής Κυρώσεων. όπως επίσης και άλλες θέσεις στο Διεθνές Ποινικό για την α, ε, ε, τέος Δεν τα πέτυχα όλα, ίσως τα πιο πολλά. Έχουμε επίσης τον κύριο Κάτινγκ, είναι ο Γενικό Γραμματέα των Κοινοβουλευτικών για Παγκόσμια Δράση. Τα τελευταία 13 χρόνια ο κύριος Κάτιν προώθησε την καθολικότητα και την αποτελεσματικότητα των διεθνών ποινικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από 100 περίπου χώρες με τη δική του βοήθεια και με τη δική του συνεργασία υπήρξε επικύρωση του καθεστώτος λειτουργίας, του κανονισμού λειτουργίας 56, από 56 από τις 124 χώρες που συμμετέχουν. Συμμετοχή στην δημιουργία λοιπόν της Διεθνούς Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης και του Τεράμου στην Ιταλία. Έχουμε επίσης μαζί μας σήμερα τον κύριο Μπαρίκα, υπεύθυνο της μόνιμης εθνικής αντιπροσωπίας του Λίχτενστάιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μπαρίκα έχει εκπροσωπήσει το Λίχτενστάιν σε πολλές διεθνείς υποθέσεις σχετικές με το ποινικό δίκαιο και τις διεθνείς σχέσεις μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, ήταν επίσης σύμβουλος του Προέδρου των Διαπραγματεύσεων που οδήγησε στην υιοθέτηση των τροπολογιών του ε, Διεθνούς Ποινικού, του Κανονισμού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Βιέννης και πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Κολονίας. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Πρόστα, όχι παραπάνω από 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να ασχοληθούμε με τα θέματα της ατιμορρησίας και τον ρόλο του διεθνούς ποινικού. Γνωρίζω ότι θα υπάρξει ειδική, αν θέλετε, αναφορά στο έγκλημα της επίθεσης αυτής ε, θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο των εργασιών του δικαστηρίου στην παρούσα φάση και ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει. Η κεντρική ο πυρήνας της εντολής ε, του ε, δικαστηρίου αυτού ασχολείται με θέματα γενοκτονίας και με ε, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τώρα προστίθεται και το θέμα του εγκλήματος της επιθέσεως. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι το δικαστήριο έχει πολλή δουλειά με την κομβική του αν θέλετε εντολή δίωξη των εγκλημάτων αυτών. Η εισαγγελία, ε, ένα όργανο φυσικά του Διεθνούς Δικαστηρίου και διεξάγει στην παρούσα φάση 10 ανακριτικές διαδικασίες για την Ουγκάντα, την Δημοκρατία του Κονγκό, το Ντάρφουρ, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν δηλαδή, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Κένια, τη Λιβύη, την Ακτή του Ελεφαντοστού, το Μάλι και την Γεωργία. Εννέα είπα, αλλά υπάρχουν δύο διαφορετικές έρευνες για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Είναι σημαντικό σχετικά με τα σχόλια τα οποία θα κάνω αργότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την Αφρική να γνωρίζουμε από τις δέκα αυτές καταστάσεις με τις οποίες ασχολείται η εισαγγελία. Πέντε από αυτές αναφέρθηκαν ή μάλλον έφτασαν στο δικαστήριο από τις ίδιες τις χώρες τις οποίες αφορά. Σε δύο περιπτώσεις υπήρξε κατάθεση του φακέλου από το Συμβούλιο Ασφαλείας και υπάρχουν τρεις ε, περιπτώσεις τις οποίες ε, η ίδια η εισαγγελία επέλεξε προς ε, έρευνα Γεωργία, Κένια και ακτή του Ελεφαντόδοντος. Έχουν υπάρξει δέκα προκαταρκτικές διαδικασίες σε διάφορες περιοχές του κόσμου όπως Μπουρούντι, Αφγανιστάν, Κολομβία, Γκαμπόν, Γουινέα, Ιράκ σχετικά με τα Βρετανικά στρατεύματα, Νιγηρία, Παλαιστίνη, ε, σκάφη ε, τα οποία ανήκουν στα νιολόγια της ε, Καμπότζης, της Ελλάδας και της Ουκρανίας. Στο δικαστήριο λοιπόν, στην έδρα του δικαστηρίου συζητώνται υποθέσεις. Πέρυσι ήταν ένας πολύ απαιτητικός χρόνος για το διεθνές ποινικό. Εκδόθηκαν τρεις αποφάσεις, η μία είναι τελική Επτά καταδίκες ανακοινώθηκαν και αυτό θα έλεγα στην ουσία καλύπτει νέα εδάφη ε, σε σχέση με τη δικαιοδοσία. Είχαμε επίσης και την πρώτη φορά που κάποιος δήλωσε ένοχος και είχαμε και την πρώτη καταδίκη σχετικά ε, με την καταστροφή πολιτιστικών μνημείων στο Τιμπουκτού. Επίσης υπήρξαν, ε, ε, ε, σε, υπήρξε σεξουαλική βία, ανάληψη ευθύνης άσκηση βίας και υπήρξαν επίσης και παρεμβάσεις στην διαδικασία της δικαιοσύνης. Απειλές σε μάρτυρες και βία εις βάρος μαρτύρων. Πέρυσι ασχοληθήκαμε λοιπόν με τρία θέματα ταυτόχρονα στο δικαστήριο σχετικά με, το, με την ακτή του ελεφαντόδοντος, με την Ουγκάντα και επίσης ε, πάντη στην Ουγκάντα με τον στρατό αντίστασης του Θεού όπως λέγεται, το Lord Resistance Army. Εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα της προσθήκης της τροπολογίας και το θέμα της δυνατότητας αποζημίωσης των θυμάτων όταν αναγνωρίζεται η βία εις βάρος τους. Υπάρχουν και δύο εφέσεις που βρίσκονται στο τελικό στάδιο σχετικά με αποφάσεις ε, οι οποίες έχουν εκδοθεί και υπάρχουν επίσης ε, και συζητήσεις εξοδικαστικές γύρω από πιθανές αποζημιώσεις. Υπάρχουν λοιπόν ε, πάρα πολλές ενδιαφέρουσες υποθέσεις. Εγώ θα μπορούσα να συζητήσω πολλά από τα θέματα αυτά προς το δικό σας όφελος, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Κάποιες από αυτές είναι εσωτερικές και τις ελέγχει το δικαστήριο και κάποιες άλλες είναι εκτός της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου. Ένα από τα θέματα τα οποία τίθενται, ε, θα έλεγα γενικά, στην ε, διεθνή δικαιοδοσία είναι ο σύνδεσμος του χρόνου με τον οποίο διεξάγονται οι διαδικασίες αυτές και της αποδοτικότητας του της διεθνούς δικαιοσύνης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πολύ κριτική εις βάρος του δικαστηρίου. Υπάρχει κριτική και υπάρχουν ανησυχίες τις οποίες έχουμε λάβει υπόψη, έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου έχει προσπαθήσει σαν βασικό στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του δικαστηρίου. Οι δικαστές έχουν εισαγάγει συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ήδη έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τον χρονισμό τον οποίο ακολουθούμε σαν δικαστήριο για να πάρουμε αποφάσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο άπτεται συνεπώς της αποτελεσματικότητας του διεθνούς ποινικού. Πάντως η κριτική και οι προκλήσεις τις οποίες θα έχετε σίγουρα ακούσει μέχρι τώρα είναι κυρίως αυτές οι οποίες προέρχονται από το λεγόμενο εξωτερικό πλαίσιο. Σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στο δικαστήριο και την Αφρική. Έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη κριτική εις βάρος του δικαστηρίου ότι ασχολούμεθα κυρίως μετά της Αφρικής και ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στην Αφρική. Ταυτόχρονα, το φθινόπωρο υπήρξαν τρεις χώρες της Αφρικής που αποχώρησαν από τη Συμφωνία της Ρώμης, αλλά η κατάσταση αυτή, και χαίρομαι που σας δίνω περισσότερες πληροφορίες αργότερα γι' αυτό, είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα έλεγα, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο η Αφρική ήταν μία από τις περιοχές οι οποίες συνεισέφεραν τα μάλλα στην δημιουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Είναι προφανές λοιπόν ότι είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή ομάδα και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην Αφρική. Ε, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλές ε, χώρες οι οποίες ε, παρενέβησαν, θα έλεγα προσέφυγαν μόνες τους στο δικαστήριο. Ήταν αυτοαναφορικές δηλαδή οι παρουσιάσεις τις οποίες έκαναν των θεμάτων τους. Ιδιαίτερα εκεί όπου είχαν προηγηθεί στο παρελθόν συγκρόσεις. Υπάρχει και άλλο ένα σημαντικό θέμα το οποίο εξηγεί το γιατί υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις, είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο συγκυριακό πλαίσιο γύρω από τα θέματα της Αφρικής. Η Αφρική λοιπόν συνεχίζει την προσπάθεια, ή μάλλον το δικαστήριο συνεχίζει την προσπάθεια την οποία κάνουμε. τώρα οι δύο αιτήσει αποχώρησης ακύρωσαν την αποχώρησή τους η Νότια Αφρική και η Γκάμπια επίσης έκανε το ίδιο πράγμα μετά από την αλλαγή της κυβέρνησης στη συγκεκριμένη χώρα. Υπάρχει η ανακοίνωση της αποχώρησης του Μπουρούντι η οποία θα γίνει ένα χρόνο μετά από την κατάθεση του φακέλου αλλά από τότε δεν έχουν υπάρξει άλλες αποχωρήσεις παρά το ότι είχε θεωρηθεί αυτό ότι θα δημιουργούσε μια πλημμυρίδα αποχωρήσεων. Υπήρξαν ε, λοιπόν πάρα πολλές δυσκολίες ε, για το δικαστήριο και από την Αφρική αλλά και γενικότερα γιατί σαν παραδείγμα το δικαστήριο ασχολείται με συγκεκριμένες περιοχές. Ήταν μια συγκεκριμένη ερώτηση ε, για συγκρούσεις και σε άλλες περιοχές όπως η κατάσταση στην Συρία γιατί το δικαστήριο δεν έχει ασχοληθεί με τα τι συμβαίνουν εκεί. Ο λόγος είναι ε, ότι δεν εξαρτάται από το διεθνές ποινικό. Εμείς βασιζόμαστε σε μια συγκεκριμένη συνθήκη και γι' αυτό η δικαιοδοσία μας είναι περιορισμένη στις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στις 124 αυτές χώρες. Και αυτές οι 124 χώρες θα πρέπει να εμπλέκονται σε μια τέτοια κατάσταση, είτε άμεσα σε σχέση με το έδαφος τους το ίδιο δηλαδή, είτε ή η υποτεθέμενη εμπλοκή να αφορά πολίτες της συγκεκριμένης χώρας. Συνεπώς λοιπόν ο κανονισμός της Ρώμης δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία και διεθνή εφαρμογή και συνεπώς η δικαιοδοσία του δικαστηρίου δεν καλύπτει περιπτώσεις σαν της Συρίας. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό όταν βλέπουμε τέτοιου είδους σειράξεις. Η μοναδική λύση για ένα τέτοιο πρόβλημα είναι να υπάρξουν περισσότερες χώρες και να επιδιωχθεί ο καθολικός χαρακτήρας. Αυτό είναι ζωτικό για την αξιοπιστία του δικαστηρίου. Είναι σημαντικό επίσης διότι η η εφαρμογή αν θέλετε του καθεστώτος της Ρώμης είναι κάτι το οποίο βασίζεται στην έννοια της αλληλεγγύης και στήριξης των θυμάτων. Είναι μια βασική προτεραιότητα για το δικαστήριο και μια προτεραιότητα την οποία επιδιώκουμε στα πλαίσια του στόχου του καθολικού χαρακτήρα των αποφάσεων. Εγώ είπα ότι συνεργαζόμαστε επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλα διεθνή όργανα Είμαστε ευγνώμονες για την ενίσχυση την οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δικαστήριό μας και σε λειτουργικό επίπεδο και σε επίπεδο συνεργασίας και σε επίπεδο πολιτικής στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο έχει υιοθετήσει πάρα πολλά ψηφίσματα υποστηρίζοντας τη λειτουργία μας. Αυτό είναι κάτι το σημαντικό λοιπόν για τις εργασίες του δικαστηρίου μας και εκτιμάμε δεόντως τις αλληλοεπιδράσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία θα μπορούσα να σταθώ, αλλά θα περάσω τον λόγο στους συναδέλφους που θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις και σχόλια. Thank you so much. We give the... Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κατίν, για 10 λεπτά παρακαλώ. Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία που έχω να βρίσκομαι ενώπιό σας και τιμή μου που ε, ως ε, Ιταλός βρίσκομαι στην αίθουσα που φέρει το όνομα του Αλτσίντε Ντεκάσπερη. Θέλω να αποτίσω και ένα φόρο τιμής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και η δικαστής πρόστα. Ήταν ε, πρωτοπόρο στη διεθνή ποινική δικαιοσύνη. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζήτησε ένα διαρκές δικαστήριο, ε, ενώ ήταν περιπλανόμενη και πλανόδια δικαιοσύνη στη Ιουκοσλαβία και αλλού για τις γενοκτονίες ad hoc κάθε φορά ε, δημιουργήθηκαν δικαστήρια. Από σήμερα 24.000 και παραπάνω θύματα από την Αφρική ζήτησαν ε, να συμμετέχουν σε διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου. Πάνω από 10.000 έχουν αναγνωριστεί ε, ως συμμετέχοντες στις δίκες. 6.000 Γεωργιανοί επίσης ζήτησαν να εμφανιστούν ενώπιον το δικαστηρίο. δηλαδή πάνω από 30.000 Χιλιάδες έχουν έρθει στη Χάη. Αυτό είναι Ε, πολύ σημαντικό για το δικαστήριο. Ενώ η αντίθεση και η αντίσταση ε, προς το δικαστήριο έρχεται κυρίως από ηγέτες, από εκείνους που θεωρούν ότι είναι υπεράνω του νόμου ε, και δεν είναι ικανοποιημένοι με την έννοια ότι υπάρχει στη Χάγη ένα διεθνές δικαστήριο που ενδεχομένως να τους αφορά και να γεμίσει αυτό το κανό ατιμορρησίας που μπορεί να υπάρχει στην εθνική δικαιοσύνη. Ε, για τις ε, φρικαλαιότητες και τα εγκλήματα που ε, διαπράττονται. Το Διεθνές λοιπόν ποινικό δικαστήριο είναι για μας πολύ σημαντικό θεσμός και ακριβώς επειδή ανταποκρίνεται στο ρόλο του δημιουργεί εντάσεις και αντιπαλότητες. Στην Αφρική δεν έχει αντιπάλους γιατί λειτουργεί με σωστό τρόπο. Και αυτή είναι η φυσική αντίδραση ορισμένων ηθινόντων που πολλές φορές μπορεί να είναι πρόεδροι κρατών που θέλουν να συνεχίσουν ατιμόρυτοι να ακολουθούν την τακτική τους. Αλλά τώρα μπορεί να τους εκδοθεί ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης και να παραπευθούν στο διεθνές ποινικό δικαστήριο, αλλά αυτό τους περιορίζει ε, την ασυδοσία τους. Σήμερα είναι μαζικά τα εγκλήματα που διαπράττονται σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου και εξαιρούνται από την δικαιοδοσία ε, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η Συρία, για παράδειγμα, που είναι μακράν η ε, πιο αιματηρή σύγκρουση και σύραξη στον κόσμο. Εμείς, ε, βουλευτές για την παγκόσμια δράση και όλες οι μήκοι όπου εντάσσονται σε αυτό το φάσμα, όπως Human Rights Watch και η Διεθνής Αμνηστία, Είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε συμφωνία ε, ή συνεννόηση για τιμωρησία ε, που υπονομεύει και παρεμποδίζει το έργο του Διεθνούς Πυρηνικού Δικαστηρίου. Αυτό το είδαμε με σάρκα και οστά στο Συμβούλιο Ασφαλείας το 2014 το Μάιο με το ΒΕΤΟ ε, με τη Μοσούλη πριν πέσει στα χέρια του ISIS, όπου η Κίνα και η Ρωσία έβαλαν βέτο σε μια πρόταση της Γαλλίας που την υποστήριζαν όλα τα υπόλοιπα κράτη ε, μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να παραβευθεί η Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Για να δημιουργηθεί μια ζώνη ατιμωρησίας στη Συρία. Και υπάρχουν και άλλες πολύ σοβαρές καταστάσεις σειράξεων με μαζικές φρικαλαιότητες. Βλέπε η εμένη που δεν βλέπει τόσο πολύ το φως ε, της δημοσιότητας η κατάσταση αυτή. Γίνονται διάφορες συνεννοήσεις για να συγκαλύπτονται τα εγκλήματα που διαπράττονται εκεί. Άρα υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα σήμερα τιμωρησία στον κόσμο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις όλα αυτά συμβαίνουν εκτός της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και είναι προς τιμή του δικαστηρίου ότι έχει αντίκτυπο. Έχουμε συλλέξει από τα μέλη μας μαρτυρίες και ποιος, μία από τις πιο συγκινητικές ήταν κάτι που συνέβη στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, όπου η αντιπολίτευση είχε ορίσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία στην Κινσάσα να είναι νεκρή πόλη. Δηλαδή, σταματήσουν τα πάντα και ενώταν μεγάλη διαμαρτυρία και συγκρούσεις ε, αντιφρονούντων με την κυβέρνηση. Μας, μας ζήτησαν να δούμε βουλευτές ε, από διάφορα κόμματα του πολιτικού φάσματος και προσκαλέσαμε ε, διαφόρους πολιτικούς και έμαθαν ότι η εισαγγελία είχε φτάσει στην Κινσάσα και δεν υπήρξε το παραμικρό. Ε, επεισόδιο. Ακριβώς επειδή ήταν παρόν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ορατό. Ουσιαστικά δεν, μπορεί κανείς να ποσοτικοποιήσει κάτι που δεν συμβαίνει. Αλλά ξέρουμε ότι από τις αποφάσεις εμποδίζονται ορισμένε αρνητικές εξελίξεις και ε, ε φρικαλαιότητες για ε, τομεί και γεωγραφικές περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Βέβαια αυτό δεν είναι πανάκια, ε, ούτε ε, τις αιματηρές συγκρούσεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ούτε την οδυνερή και ματηρή μετάβαση της εξουσίας ή του καθεστώτος όπως συμβαίνει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Οι μασικές φρικαλαιότητες είναι εγκλήματα που διαπράττουν συνήθως ηγέτες ηγέτες που έχουν στα χέρια τους τον κρατικό μηχανισμό ή και μη κρατικούς ε, παράγοντες και φορείς που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεγάλες ε, στρατιωτικές επιθέσεις που κυρίως τρέφονται κατά του άμαχου πληθυσμού. Στην Ιρεμβέργη το 1945 αναγνωρίσαμε τέσσερα διεθνή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, του που το 1948 ε, έγινε σύμβαση, τα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ειρήνης. Τα εγκλήματα κατά της ειρήνης εξαιρέθηκαν ή δεν θεωρούν δεν θεωρείται ότι ήταν ενεργό τμήμα της δικαιοδοσίας στη δεκαετία του 1990, γιατί όλα αυτά θεωρούν το ζητήματα εσωτερικής σύραξης και όχι διεθνούς το 98 όταν εγκρίθηκε το καταστατικό της Ρώμης και θυμάμαι το δικαστή Hans Peter Gauck εδώ στο Κοινοβούλιο πριν μερικά χρόνια ε, πριν αποβιώσει δυστυχώς ε, καταφέραμε στο άρθρο 5 του καταστατικού της Ρώμης να εντάξουμε και το έγκλημα της επίθεσης που θα έπρεπε να επανέλθει ακριβώς εκεί που είχε ενταχθεί το 1945 και ερχόμαστε τώρα το 2017 με 34, 35 κυρώσεις μάλιστα, γιατί η Αργεντινή πρόσφατα, καλά, 34 γιατί με την Πορτογαλία και την Αργεντινή επίκυνται διάφορες εξέλιξεις. Ας μην προτρέχουμε εμείς ε, το γεγονό και θα πρέπει να δούμε ε, ε, κατά πόσο ενεργοποιείται αυτό το έγκλημα στις 17 Ιουλίου του 2014 μετά από πρωτοβουλία, πρωτοβουλία της κυρίας Λοχμπίλερ εγκρίθηκε ομόφωνα ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν δεν απατώμε ένας μόνο ψήφισε κατά και στο ψήφισμα αυτό απευθυνόταν μια έκκληση για την υποστήριξη της ε, Καμπάλα, των τροπολογιών Καμπάλα. Αυτή είναι η θετική πλευρά, αλλά σε κάθε περίπτωση που είναι συμβιβασμό υπάρχει και η ανετική πλευρά. Οι επιθέσεις που αναφέρατε εσείς Πρόεδρε στην αρχή το δικαίωμα της επίθεσης όπως αναφέρεται στο ψήφισμα 3314 του 1974 ε, είναι περιορισμένο, διότι υπάρχει παράγραφος 1 που μας λέει ότι το έγκλημα της επίθεσης συντελείται μόνο όταν ένας ηγέτης στρατιωτικός ή πολιτικός παρανόμος ε, προβαίνει σε μια επίθεση κατά άλλης χώρας που λόγω του χαρακτήρα, του ειδικού βάρους και της κλίμακας παραβιάζει το χάρτη θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων του ΙΕ. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει με, το μέγεθος, με την κλίμακα, με το χαρακτήρα και περιορίζει την... Επειδή μάλλον ορίζει το τι εστί η επίθεση για να μην υπάρχουν γκρίζε ζώνες. Γιατί ε, δεν είναι μόνο τόσα συνέβησαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ή σε άλλου πολέμου. Για να μπορέσει ο συμβασμό να γίνει δεκτό από όλου. Και όντω έγινε δεκτό, διότι εγκρίθηκε συνενετικά. Ε, ακόμα γίνονται συζητήσεις για το πώς ε, ερμηνεύουμε το πότε ενεργοποιείται, το πότε τίθεται σε ισχύ. Αυτά είναι τεχνικά ζητήματα, αλλά η δική μου οργάνωση, οι βουλευτές για την ε, παγκόσμια δράση, συμφωνεί με όλα αυτά η ισότητα όλων απέναντι στον νόμο είναι τα ίδια τα θεμέλια του συστήματος καταστατικού της Ρώμης. Τελειώνω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ακόμα να κάνει τη διαφορά και στο παρελθόν το έπραξε. Είναι η μόνη περιφαρειακή οργάνωση, ένας διεθνή οργανισμός με πρόγραμμα δράσης, με κοινή θέση που σημαίνει δραστηριότητες επιτόπου με πολιτικές ρήτρες όπως το άρθρο 97 της Συμφωνίας του Κοτονού κτλ. Αλλά θα ήθελα να σας φέρω το εξή μόνο για να είμαι ακριβής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο στεναρή. Έδειξε στένος και πυγμή στο παρελθόν, αλλά ακόμα περισσότερο στη συνεργασία με την Ουκρανία, έτσι ώστε να προσχωρήσει σε κάτι που συμφώνησε το Κοινοβούλιο και ενέκρινε και κυρώθηκε στη Συμφωνία Σύνδεσης. Είναι μια χώρα από την οποία έχει προσαρτήσει παράνομα επικράτεια ένα άλλο κράτος. Βέβαια, το έγκλημα της επίθεσης ε, τίθεται σε ισχύ τέλη του 2017. Ε, δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν έχει ισχύ, δεν επηρεάζει πρόσωπα που είναι πολίτες κράτους μη ε, μέλους. Όποιος όμως χρησιμοποιεί τη βία παράνομα και ε, προβαίνει σε εγκλήματα πολέμου ή κατά της ανθρωπότητας μπορεί να θεωρηθεί επιφαρυντικό στοιχείο από τους ε, δικαστές. Καλό λοιπόν, απευθύνω έκκληση και πάλι προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το ζητήσει αυτό, να ζητήσει από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να υψώσει την ε, φωνή της προς τους Ουκρανούς εταίρους άλλαξαν το Σύνταγμα αλλά δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει αυτή την πρόταση και θα τους βοηθούσε ενδεχομένως σε μια πίεση από τους ε, εταίρους τους. Και να περάσουμε τώρα στο τρίτο μιλητή, στον κύριο Μπαρίγκα, για 10 λεπτά. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα και είναι και πρόκληση να μιλήσω μετά από αυτούς τους δύο εγνωσμένου κύρους ομιλητές, οι οποίοι σας παρουσίασαν μια αρκετά πλήρη εικόνα ήδη. Αυτό που θα μπορούσα να δω, ίσως να, σας, να κάνω, ίσως να σας δώσω λίγο περισσότερο το το ιστορικό του εγκλήματος της επίθεσης και να σας πω και δύο λόγια ίσως για την νομική και πολιτική σημασία της μελλοντική ενεργοποίησης της δικαιοδοσίας του ποινικού δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης. Ως προς το ιστορικό, όπως ε, ανέφερε ήδη ο Ντέιβιτ, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από τις ε, δίκες του Ισνιρεμβέργη και του Τόκιο μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, Ιαπωνέζοι ηγέτες και οι ηγέτες ε, της ναζιστικής Γερμανίας καταδικάστηκαν για τα λεγόμενα εγκλήματα κατά της ειρήνης και ο όρος έγκλημα της επίθεσης και έγκλημα κατά της ειρήνη θα μπορούσαν ίσως να θεωρηθούν συνώνυμοι. Πιο συγκεκριμένα, τότε αυτοί οι άνθρωποι καταδικάστηκαν για το σχεδιασμό, προετοιμασία, ε, την παρακίνηση ε, μιας, ενός επιθετικού πολέμου. Αλλά ε, τότε δεν είχε διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο επίθεση. Και αργότερα η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών χρειάστηκε αρκετές δεκαετίες για να ορίσει τι ακριβώς σημαίνει επίθεση. Και με τον όρο επίθεση θα πρέπει να κάνουμε διάκριση αυτού που περιλαμβάνεται στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, όπου ορίζεται ως η απαγόρευση της ε, χρήσης βίας, ενώ το έγκριμα της επίθεσης είναι κάτι πέραν αυτού, έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και είναι κάτι πολύ πιο ε, ουσιαστικό. Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών λοιπόν συμφώνησε μετά από δεκαετίες ε, για τον ορισμό της επίθεσης, ο οποίος ε, ξεκίνησε από το άρθρο 2.4 για τον ορισμό της χρήσης της βίας και ε, αυτό νομίζω ότι έχετε να προσθεθεί και σε αυτό που είπε προηγουμένως ο πρόεδρο. Αναφέρθηκε σε διάφορα εγκλήματα, εισβολή, βομβαρδισμό κλπ. Για να θεωρηθούν αυτέ οι πράξει εγκλήματα θα πρέπει να είσαι κατά παράβαση τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, που σημαίνει ότι δεν θα γίνεται λόγω άμυνας, λόγω αυτοάμυνας ή δεν θα υπάρχει έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπήρχε λοιπόν το 1974 ορισμός ε, για το τι ακριβώς σημαίνει επίθεση από ένα κράτος κατά ενός κάποιου άλλου. Αλλά ε, δεν υπήρχε ορισμός για το τι σημαίνει το έγκλημα για αυτόν ο οποίος βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου κατηγορούμενος. Για να γίνει αυτό έπρεπε να φτάσουμε στη διάσκεψη της Ρώμης του 1998 που όπως ο Ντέιβιτ ανέφερε οι αντιπροσωπείες κατάφεραν τουλάχιστον να έχουν ε, κάτι, μία μνήα, κάτι παραπάνω ίσως από την μνήα στην, ε, στο καταστατικό της Ρώμης. Το καταστατικό της Ρώμης λέει ότι τα συμβαλώμενα μέρη στο καταστατικό δέχονται τον ορισμό μεταξύ άλλων και του ορισμού της επίθεσης. Παρά το γεγονός ότι τότε δεν υπήρχε σαφής αναφορά στο καταστατικό της Ρώμης και τότε αυτό το οποίο αποφασίστηκε ήταν να δοθεί εντολή για να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση η οποία θα οδηγούσε στον ορισμό και θα είχαμε και περισσότερη σαφήνεια για το ε, τι δικαιοδοσία έχει το δικαστήριο. Αυτά συνέβησαν μεταξύ του 2003 και του 2010 και πρόεδρος ήταν ο πρέσβης του Λίχτενστάιν των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και ίσως και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εγώ εδώ σήμερα και θα μπορούσα ιδιαίτερα στις ερωτήσεις και απαντήσεις αργότερα να σας πω και λίγα περισσότερα για το τι συνέβη στη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Για να συνοψίσω, ε, εκείνη την επταετία βρήκαμε ε, ε, δυνατότητα να συμφωνήσουμε σε δύο τμήματα των τροπολογιών Καμπάλα. Το πρώτο ήταν ο ορισμός της επίθεσης, το οποίο αναφέρθηκε ήδη αρκετές φορές σήμερα. Αναφερόμαστε στις πιο σοβαρές μορφές παράνομης χρήσης βίας, όπως προβλέπεται από τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και αυτό βρέθηκε το Φεβρουάριο του 2009, ένα χρόνο πριν από την επίσημη διάσκεψη της Καμπάλα, που σημαίνει ότι ο ορισμός αυτός καθεαυτός δεν αποτελεί επίμαχο ζήτημα και πρέπει να πω ότι τότε εγκρίθηκε όχι μόνο από τα συμβαλόμενα μέρη του ποινικού δικαστηρίου, αλλά ο ορισμός εγκρίθηκε σε μια ομάδα εργασίας η οποία ήταν ανοιχτή σε όλα τα ε, κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Είτε συμμετέχουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είτε όχι, μπορούσαν να ε, ε, έρθουν σε αυτή την ομάδα εργασίας και να αποδεχτούν τον ορισμό. Η δεύτερη στήλη αυτής της δέσμης μέτρων ήταν ε, το θέμα των όρων της δικαιοδοσίας. Μπορεί να σας φαίνεται τεχνικός αυτός ο όρος, αλλά εδώ υφέρουν τουλάχιστον δύο ομάδες προβλημάτων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ακαθόδη. Το πρώτο είναι ποιος θα πρέπει να είναι ο, ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ε, επιβολή, την ε, ε, εκδίκαση ε, εγκλημάτων επίθεσης του ποινικού δικαστηρίου στη συνέχεια. Εκεί βρήκαμε ένα αξιοσημείωτο συμβιβασμό, δηλαδή ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν θα εξαρτάται από πρώτερη συγκατάθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας για να κάνει έρευνα για το έγκλημα της επίθεσης. Υπάρχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σε αυτή την περίπτωση, αλλά κατ' ουσίαν καταφέραμε να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία του ποινικού δικαστηρίου ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας για το έγκλημα της επίθεσης. Ε, το δεύτερο τμήμα τη δέσμη μέτρων για τη δικαιοδοσία ήταν το θέμα τη ε, συγκατάθεση. Σε ποιο βαθμό ε, θα πρέπει να περιορίζεται η δικαιοδοσία του ποινικού δικαστηρίου για να συμπεριλάβουν κράτη τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν συμφωνήσει για τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό για το καθεστώς του ποινικού δικαστηρίου ε, για τα υπόλοιπα τρία βασικά εγκλήματα δεν χρειάζεται συγκατάθεση όλων των ενδιαφερομένων κρατών. Εάν υπήκος ε, κράτους που δεν είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού διαπράξει ένα έγκλημα στο Διεθνές Ποινικό, ε, σε χώρα που είναι μέλος του Ποινικού Δικαστηρίου υπάρχει δικαιοδοσία παρά το γεγονός ότι ε, δεν συμμετέχει συγκεκριμένη χώρα. Εκεί υπήρχε διάσταση απόψεων βέβαια για το κατά πόσον θα πρέπει να ισχύει το ίδιο σύστημα και για το έκλειμα τη επίθεση. Κάποιε χώρε ήθελαν να διατηρήσουν ακριβώ το ίδιο σύστημα, το οποίο είναι καλό για πιθανά θύματα, του παρέχει προστασία ε, γιατί αν η χώρα αυτή κυρώσει τις τροπολογίες και ακόμα και αν ένα ε, κράτος που δεν είναι μέλος του ποινικού δικαστηρίου διαπράξει έγκλημα σε κράτος που είναι, υπάρχει δικαιοδοσία, αλλά κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό υπερβαίνει τα όρια ε, και ήθελαν κάτι πιο παραδοσιακό που δεν βασίζεται στη συγκατάθεση και επέμεναν να υπάρχει κάτι στο οποίο θα χρειάζεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο συγκατάθεση και όλων των κρατών που εμπλέκονται και ε, τελικά έπρεπε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό και καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό που περιορίζει βέβαια αρκετά τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης ε, και βασίζεται στη συγκατάθεση. Και το σύστημα αυτό το οποίο βασίζεται στη συγκατάθεση σημαίνει ότι αφενός αποκλείονται επιθέσεις οι οποίες διαπράττονται από χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν ε, δηλαδή χώρες που δεν συμμετέχουν στην δικαιοδοσία είτε ως θύματα είτε ως θήτες δεν ε, συμμετέχουν και ε, επίσης υπάρχει δυνατότητα opt-out. Δηλαδή υπάρχει το τεκμήριο ότι έχουν αποδεχτεί την ε, δικαιοδοσία αλλά μπορούν να κάνουν δήλωση και να επιλέξουν να μην συμμετέχουν opt λοιπόν. Και εδώ υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο χρειάστηκε να συμπεριλάβουμε στο πακέτο στην Καμπάλα, Ένα ειδικό μηχανισμός ενεργοποίησης, κάτι το οποίο είναι αρκετά παράδοξο, αλλά αντικατοπτρίζει το πόσο περίπλοκος ήταν αυτός ο συμβιβασμός. Οι χώρες δεν ήθελαν να ξεκινήσει η ισχύ του αμέσως, ήθελαν λίγο περιθώριο σε αυτή τη σύνθετη λύση και είπαν ότι έχουμε δύο λύσεις για να ασκήσει το δικαστήριο την δικαιοδοσία του. Καταρχάς θα θέλαμε τουλάχιστον 30 κυρώσεις για να δείξουμε ότι υπάρχει πολιτική υποστήριξη για τις τροπολογίες και θα θέλαμε απόφαση από τα συμβαλώμενα μέρη Δηλαδή να ανοίξει ο διακόπτης και να ενεργοποιήσουμε αυτές τις τροπολογίες και αυτό φυσικά ε, δεν μπορεί να γίνει πριν από το 2017. Είμαστε στο 2017, οι συζητήσεις συνεχίζουμε και περιμένουμε απόφαση το Δεκέμβριο του τρέχοντος. Όσον αφορά τις κυρώσεις, ε, πρέπει να πω ότι έχουμε 34 κυρώσεις μέχρι σήμερα και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Ε, να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε στο μεταξύ. 18 κράτη-μέλη έχουν κυρώσει τις τροπολογίες και ελπίζουμε ε, να συμμετέχουν ε, ακόμα περισσότερα. Και επίσης, όπως είπε και ο Ντέιβιτ, Υπήρξαν κάποια πέρα δόθε όσον αφορά κάποιες τεχνικές πτυχές, το μηχανισμό του opt-out, τον οποίο θα μπορούσα ίσως να σας αναπτύξω λίγο περισσότερο στη διάρκεια των ερωτήσεων για να ολοκληρώσω τρει σύντομε παρατηρήσει για τη σημασία των τροπολογιών Καμπάλα. Πρώτον, οι τροπολογίε Καμπάλα ολοκληρώνουν ένα πολύ μεγάλο κενό στο διεθνέ ποινικό δίκαιο. Το έγκλημα της επίθεσης δεν έχει ε, τύχη καταδίκης από τη δίκη της Νιρεμβέργης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι τι σημαίνει να επιτρέψουμε στο δικαστήριο να καταδικάζει για το έγκλημα της επίθεσης. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπουμε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εφαρμόσει την πιο σημαντική διάταξη της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα εφαρμόζει την απαγόρευση της παράνομης χρήσης βίας στις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Δεύτερον, θα υπάρχουν πολλέ περιπτώσεις ενώπιον του δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης και με αυτό ολοκληρώνω ε, απίθανο γιατί είναι πολύ περιορισμένη η δικαιοδοσία, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την εκδίκαση του εγκλήματος της επίθεσης από πλευράς ποινικού δικαστηρίου και το ανέφερε και η κυρία Πρόστ, είπε ότι είναι πολύ απασχολημένο το δικαστήριο και έχει πολλή δουλειά. Μπορεί το έγκλημα της επίθεσης να ε, προσθέσει δουλειά στο δικαστήριο, αλλά συνήθως μπορεί να συμβεί το αντίθετο. Συνήθως δεν διαπράτεται μόνο ένα έγκλημα, αλλά πολλαπλά εγκλήματα. Και το έγκλημα της επίθεσης είναι ε, αρκετά αρκετά εύκολο στην εκδίκασή του, διότι είναι το έγκλημα το οποίο διαπράττει ο ηγέτης. Είναι πολύ πιο εύκολο να αποδείξουμε ότι ένας ηγέτης είχε σκοπό να επιτεθεί σε μια χώρα από το να αποδείξουμε ότι είχε πρόθεση να διαπράξουν εγκλήματα πολέμου οι στρατιώτες του εν καιρό πολέμου. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει το έγκλημα της επίθεσης και αυτό δεν το λέω ελαφρά την καρδία, είναι πιο εύκολο. Ε, και ε, τρίτον, ε, η καταδίκη είναι σε εγχώριο επίπεδο. Και πριν από την Καμπάλα, αλλά ιδιαίτερα μετά, τα κράτη-μέλη έχουν ποινικοποιήσει το έγκλημα της επίθεσης στα εγχώρια δικαστήρια στην ένωμη τάξη τους. Και αυτό φυσικά ε, είναι πολύ σημαντικό, διότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει περιορισμένη δικαιοδοσία και υπάρχει πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός ε, ε, τρόπος να δράσει αυτό ως ανασταλτικός παράγων, να υπάρχει δυνατότητα να δράσουμε όταν οι κυβερνήσει ή οι ηγέτε θέλουν να διαπράξουν το έγκλημα τη υπόθεση. Όσε επίθεση, όσε φορέ και να το πω, δεν αρκεί. Ε, θα ολοκληρώσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Σα ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σα. Ο πρώτο που έχει ζητήσει το λόγο είναι η κυρία Λόχ Μπίχλερ Πριν ξεκινήσω με την ερώτησή μου, θα ήθελα να πω ότι εμείς ξεκινήσαμε ε, την υπόθεση αυτή μισή ώρα νωρίτερα από ό,τι προεβλέπετο. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι επανειλημμένα, όταν προετοιμάζουμε μία έκθεση στην Επιτροπή μας για τα θέματα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, ε, δουλεύουμε με τρόπους ενίσχυσης του διεθνούς ποινικού. Οι συνάδελφοι όμως δυστυχώς επιδιώκουν να είναι παρόντες σε τρεις διαφορετικές επιτροπές και ξέρω συνάδελφο που εμπλέκεται ο οποίος θα έρθει στις ε, σε 10 λεπτά εδώ. Είναι λοιπόν περισσότερη η ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας για ερωτήσεις. Για σας κυρία Πρόστ πρώτα αφού σας ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές σας παρουσιάσεις. Θα ήθελα να μάθω με ποιο τρόπο μπορείτε να γεφυρώσετε σαν παράδειγμα την απόσταση που έχει το δικαστήριο στην Χάγη με τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται ε, και την κοινή γνώμη στις περιοχές όπου διεξάγονται τα εγκλήματα. Α, πώς μπορείτε να φτάσετε σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν ομιλούν την Αγγλική και δεν παρακολουθούν τα διεθνή νέα. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτοί οι οποίοι υποφέρουν από την κατάσταση αυτή ε, να κατανοήσουν ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι αυτοί οι οποίοι ε, διαπράττουν τα συγκεκριμένα εγκλήματα τιμωρούνται. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την αδικαιολόγητη για μένα θα έλεγα κριτική από πλευράς ε, των αφρικανικών κυβερνήσεων για τη προκατάληψη του δικαστηρίου. Είναι θετικό ότι υπάρχουν πολλές άλλες αφρικανικές κυβερνήσεις και κοινωνία των πολιτών απέριψαν την ε, αντίληψη αυτή. Παρ' όλα αυτά είναι η κατάσταση αρκετά εύθραστη, ακόμα και σήμερα. Θυμάμαι ότι εδώ και λίγα χρόνια έγιναν κάποιες προσπάθειες από το δικαστήριο να ξεκινήσει με ε, ένα γραφείο στο εσωτερικό της Αφρικανικής Ένωσης, έτσι ώστε οι αφρικανικές κυβερνήσεις να κατανοήσουν την συνέπεια της επικύρωσης ε, του κανονισμού. Νομίζω λοιπόν ότι και με μια νέα ηγεσία στην Αφρικανική Ένωση θα πρέπει να ξεκινήσετε να έχετε άμεση επαφή με τις ε, υπηρεσίες της Άντης. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν τι γίνεται με την κατάσταση των θυμάτων και του καταπιστεύματος για την αποζημίωσή τους. Και υπάρχει άλλη μια περίπτωση την οποία παρακολουθούμε προσεκτικά το θέμα των, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόσφατα περάσαμε ένα ψήφισμα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες. Διαβάζω στα μέσα ενημέρωσης ότι κάποιοι δικηγόροι προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή με το Διεθνές Ποινικό για την πιθανή εμπλοκή του Προέδρου των Φιλιππίνων στις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δεν ξέρω αν μπορείτε να μας το σχολιάσετε. Ερωτήσεις τώρα για τον κύριο Μπαρίγκα του Λίχτενστάιν. Εγώ είδα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014 και εκεί λέμε ότι πρέπει να συγχαρούμε τον Λίχτενστάιν διότι δημιούργησε ένα εγχειρίδιο για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού. Έχουμε 7 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν επικυρώσει και πέντε από τις χώρες αυτές προωθούν την διαδικασία, άλλες όχι. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή. Μετά τον Ιανουάριο του 2017 θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαρκές μόνιμο σύστημα σχετικά με το έγκλημα της επιθέσεως. Κατάλαβα καλά ότι αυτό θα ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2017, γιατί ήδη εμείς προετοιμάζουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ε, προς, το, προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι λοιπόν η πληροφορία αυτή πολύ χρήσιμη και θα την εντάξουμε στο ψήφισμά μας και αν μπορέσουμε να εργαστούμε καλύτερα. Τώρα, το Parliamentarian for Global Action ε, έχει έδρα τη Νέα Υόρκη, παρακολουθείτε και τις εργασίες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει πλέον ε, όπως παλιότερα ε, προσφυγή στο ΒΕΤΟ σε σχέση με το θέμα της προσφυγής στο διεθνές ποινικό για το έγκλημα της επίθεσης. Αλλά ποιο είναι το κλίμα στο εσωτερικό του, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχω καταλάβει ότι και στο παρελθόν ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα τα οποία έχουν για να πιέσουν προς την προσφυγή προς το δικαστήριο το διεθνές. Είδα ότι έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, τη μέση της Προεδρίας. Ελπίζω να πάρει το λόγο. Και θα ήθελα στα πλαίσια αυτού του ψηφίσματος να πω ότι από το 2014 the EU should adopt a common ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μια κοινή δράση για το έγκλημα της επίθεσης. Δεν το έχουμε όμως ολοκληρώσει αυτό ακόμα. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε πού βρισκόμαστε, έχει ήδη ξεκινήσει μια συζήτηση. Um, yes. Ναι, βεβαίω. Θα δώσουμε το λόγο στην υπηρεσία εξωτερική δράση, αν επιθυμεί να το λάβει, για να κάνει κάποια σχόλια. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι τμήματάξη στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ενώπιον σα και καλωσορίζω θερμά του ομιλητέ μα. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Μαθαίνω ότι αρχίσατε νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει. Δύο λόγια και με κίνδυνο να επαναλάβω δηλώσεις που έχουν ήδη γίνει. Θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς θεωρεί το καθεστώς της Ρώμης μέγα επίτευγμα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καθολικότητα των ανθρωπίνων αξιών είναι κάτι που και εμείς υποστηρίζουμε. Γιατί τα θύματα των εγκλημάτων αυτών ε, ε, αξίζει να δικαιώνονται και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη όπου και αν ζουν. Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την ε, υπόθεση αυτή, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές. Στόχος μας πιστεύουμε και αποστολή μας είναι να εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους λαούς και τις χώρες ε, για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας μέσω του δικαστηρίου. Το 2016 ήταν κρίσιμη χρονιά. Είδαμε να αποσύρονται κάποιες χώρες ή να ανακοινώνουν την απόσυρσή τους. Τώρα βρισκόμαστε σε διαφορετική κατάσταση. Ορισμένες χώρες έχουν αποσύρει το αίτημα απόσυρσης. Και νομίζω μόνο το Μπορούντι έχει απομείνει σήμερα. Το 2017 λοιπόν πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ διαφορετική χρονιά και ελπίζουμε και άλλες χώρες να προσχωρήσουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να αναγνωρίσουν την αρχή της καθολικότητας και της οικουμενικότητας. Πέρσι είχαμε και μια ετήσια έτσι, στρογγυλή τράπεζα ε, τα μέλη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και εκπρόσωποι του Διεθνούς Πενικού Δικαστηρίου. Αναφέρθηκατε σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα στην Αφρική. Θα έχετε και απαντήσεις στις ερωτήσεις που έγιναν οι ομιλητέ. Κατά την άποψή μας το 2016 ε, άνοιξε μια ε, ανάκριση για τη Γεωργία που δείχνει ότι το πεδίο εφαρμογή και δικαιοδοσία ουσιαστικά είναι παγκόσμιο. Ξέρουμε ότι η εισαγγελία εξετάζει προκατακτικά κάποια ζητήματα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και την Λατινική Αμερική. Και για τις Φιλιππίνες ιδιαίτερα, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέμα. Για το έγκλημα της επίθεσης, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, πολύ σύντομα. 18 από τα κράτη-μέλη μας έχουν κυρώσει. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κοινή θέση και ενιαία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η κυρίαρχη απόφαση κάθε κράτους μέλους να προσχωρήσει ή όχι. Αλλά αυτό συζητείται βέβαια σε μια ομάδα εργασία μας, μας που έχουμε στο Συμβούλιο και ασχολείται ακριβώς με αυτά τα νομικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είμαστε ακόμα στο στάδιο των συζητήσεων των συντονιστικών επαφών. 18 κράτη-μέλη έχουν κυρώσει και βεβαίως ενδιαφέρονται να πείσουν και τα υπόλοιπα. Αυτά. Σύντομα να σχολιάσω και κάποια άλλα που ακούσαμε. Ιδιαίτερα για την Νότια Αφρική που θέλησε να αποσυρθεί από το καταστατικό της Ρώμης, αλλά στο μεταξύ άλλαξε γνώμη. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν διακυβεύεται η ειρήνη, ούτε ε, εμποδίζεται κανείς προσχωρώντας το καταστατικό της Ρώμης να δρά διαμεσολαβητικά. Ε, πρόσφατα είδαμε στην Κολομβία να ε, ενδιαφέρεται για τη χώρα αυτή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και η ατιμορρησία ε, έχει πάψει να ισχύει. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις των ομιλητών. Επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ελπίζω θα έρθει και ο συνάδελφος Γκέρος για να λάβετε όλες τις ερωτήσεις πριν αρχίσετε να απαντάτε. Ε, συνήθως έτσι κάνουμε ένα-δύο πράγματα από την παρουσίασή σας και ίσως θα μπορούσατε να μου τα διευκρινίσετε. Είχα την τιμή να σπουδάσω νομική. Και φυσικά ε, γνωρίζω και τα, της ιστορίας ε, του δικαίου και τι κάναμε στη δίκη της Νιρεμβέργης και τι προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα και με ενδιαφέραν πολύ αυτά που είπατε ότι είναι πιο εύκολη η εκδίκαση του εγκλήματος της ε, επίθεσης γιατί αν πάμε πίσω στις δίκες της Νιρεμβέργης Θέλω σε γραμμές να πω ότι ναι μεν ήταν επιτυχία αλλά υπάρχει το τμήμα της απόδειξη ε, της επίθεση, ε, το οποίο ήταν ιδιαίτερα μεγάλη πρόκληση για τους δικαστές στην Ιρεμβέργη. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω. Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχουν ομοιότητες και ποια είναι η διαφορά ε, σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν τότε στην Ιρεμβέργη. Ιδιαίτερα το θέμα του πότε θεωρείται αιτιολογημένο ένα πόλεμο και πότε όχι. Διότι υπάρχουν και αποφάσει του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί να ε, μιλώ εν αγνία μου εδώ, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ένα-δυο πράγματα παραπάνω από αυτού. Και κάτι ακόμα το οποίο ε, θα ήθελα να ρωτήσω. Κάποιοι από εσά αναφερθήκατε στην Ουκρανία. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λίγα λόγια παραπάνω πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει ε, την ε, ε, διαδικασία στην Ουκρανία και τι θα θέλατε να κάνουμε εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά. Και μια τελευταία ερώτηση για τη δικαιοδοσία. Πολλά από αυτά τα πράγματα ε, θα ε, εμπίπτουν σε διαφορετική ενόμη τάξη. Κάποια θα είναι η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς λοιπόν ε, σκοπεύετε να επιλύσετε και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κι άλλο διεθνές πλήσιο και περιφερειακό ή διεθνές το οποίο να ισχύει σε άλλες περιοχές του κόσμου σε αυτή την περίπτωση βέβαια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι και πρώτα μεταξύ των χωρών τα οποία θα βρεθούν κατηγορούμενα, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στο μέλλον σε διεθνές ε, επίπεδο. Πώς ε, σκοπεύετε να λύσετε θέματα δικαιοδοσίας. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο. Έχουμε δει ε, θέματα δικαστηρίου στο Στρασβούργο και στο Λουξεμβούργο για το ποιο είναι το ε, κυρίαρχο δικαστήριο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Ε, έχουν λυθεί τα θέματα αυτά ή πώς τα βλέπετε εσείς από την πλευρά σας. Διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει ένα τρίγωνο δικαστηρίων σε συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης που θα μπορούσαν όλοι να ενδιαφέρονται για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν ξέρω αν έχει έρθει ο συνάδελφος. Δεν τον βλέπω εδώ. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε ε, και να σχολιάσετε τις πρώτες ερωτήσεις και μετά να δώσουμε το λόγο ξανά στο συνάδελφο σε δεύτερο γύρο όταν θα έρθει η συνάδελφος. Με την ίδια σειρά λοιπόν η κυρία Πρόστε αν θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ, πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Το πρώτο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε είναι κρίσιμο και πάρα πολύ κομβικό για μας. Ήταν πολλά τα διδάγματα που αποκομίσαμε για τα δικαστήρια για ε, τη Ρουάντα και την πρώην Ιουκοσλαβία. Πριν συσταθεί το δικό μας δικαστήριο. Πώς φτάνουμε στους ενδιαφερομένους επιτόπου όταν είμαστε τόσο μακριά. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για μας. Έχουμε ένα πρόβλημα ολόκληρο για τη διάδοση της δράσης μας ακριβώς για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ανάμεσα στη, και μόνο το γεωγραφικό ε, από τη Χάγη μέχρι τις ε, κοινότητες. Έχουμε γραφεία επιτόπου, όχι παντού, αλλά σε πολλές χώρες ε, που μας απασχολούν και Συνεχίζεται η παρουσία μας κατά τη διάρκεια της δίκης, ακροματικής διαδικασίας και κάποια άλλα ζητήματα. Και στο περιθώριο της δίκης αυτής καθ' αυτής έχουμε και αποστολές και από την εισαγγελία και από την πρόεδρο και από τη γραμματεία. Η δίκη που έχουμε αυτό το καιρό έχει να κάνει με τη Βόρεια Ουγγάντα και ε, το στρατό ε, αντίστασης του Θεού. Έχουμε λοιπόν παρουσία και ένα, και ένα ρόλο ε, ως παράστασης των θυμάτων στις διαδικασίες και στην ακροματική διαδικασία και αποζημιώσεων. Έχουν την ευκαιρία λοιπόν οι τοπικές κοινότητες να δηλώσουν τα θύματα και τα θύματα που θέλουν να συμμετέχουν στη δίκη. Βεβαίως είναι περιορισμένη η πορική δυνατότητες μας. Ε, ας πούμε για μετάφραση στις ε, εκάστοτε γλώσσες έχουμε δυσκολία και οικονομική. Ενδεχομένως ιστορικά να μην έχει δεθεί ιδέουσα προσοχή. Ε, θα ε, χρειαστεί στο μέλλον, ναι. εκφράζεται κάποια κριτική ε, για το γεγονό ότι εστιάζει το δικαστήριο κυρίω στην Αφρική. σα ανέφερα πολλές ε, περιπτώσει που οδήγησαν σε αυτό. Τώρα πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση αυτή. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο διάλογο με τις αφρικανικές χώρες. Ακούμε διάφορες φωνές από την Αφρική. Κοινωνία των πολιτών, ε, διάφορα κράτη έχουν διαφορετικές απόψεις Είμαστε πάντω πρόθυμοι να έχουμε διάλογο σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων, υπαλλήλων, ε, μελών του δικαστηρίου που συμμετέχουν σε διάφορες ε, εκδηλώσεις. Η πρόεδρος η ίδια του δικαστηρίου ήταν πρόσφατα στην Ουγγάντα με το καταπιστευματικό ταμείο. Συζήτησε τη κατάσταση με τους διαφόρους ενδιαφερομένους επιτόπου στη χώρα. Δηλαδή πολλά προσπαθούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις ε, ανησυχίες και τους προβληματισμούς ε, των Αφρικανών και της Αφρικής. Το θέμα του γραφείου παραμένει δύσκολο Έχουμε ένα σύνδεσμο στη Νέα Υόρκη ε, για συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και θέλουμε πάρα πολύ να ανοίξουμε γραφείο εδώ έτσι ώστε ε, να συνεργαζόμαστε περισσότερο με την Αφρικανική Ένωση, με γραφείο στην Αφρική ε, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει συμφωνήσει η Αφρικανική Ένωση ε, για την ε, κατάσταση του γραφείου. Κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία το θέτουμε αυτό το θέμα και στα σεμινάρια μας, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, να ενθαρρύνουμε όσο μπορούμε το διάλογο και αυτό το θέμα του γραφείου συνδέσμου. Το καταπίστευμα ενδιαφέρει πάρα πολύ την Πρόεδρο και το αναφέρει πάρα πολύ συχνά, είναι ένα στοιχείο του καταστατικού της Ρώμης και συνδέεται με αυτό. Βέβαια είναι εξάρτητο όργανο το οποίο ε, έχει θεσπιστεί για να ε, εκτελεί τις αποφάσεις για αποζημίωση που ε, επιδικάζονται συνήθως τους καταδικαστέντες, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε πρόσβαση, δεν βρίσκουμε τα περιουσιακά στοιχεία του ε, καταδικαστέντος, οπότε υπάρχει το καταπίστευμα αυτό και παρέχει και βοήθεια και συνδρομή, εκπροσωπεί το δικαστήριο ε, στην Ουγγάντα ας πούμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου έχουμε εκδώσει ε, εντάλματα, αλλά κατά τα άλλα η παρουσία μας δεν είναι δεδομένη, αποσιάζουμε από την περιοχή και στο καταστατικό της Ρώμης είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στο όλο σύστημα, το ταμείο, το καταπιστεύμα για να δούμε πώς βοηθούμε τα θύματα. Αγωνιζόμαστε συνεχώς για να για εξέβρεση κονδυλίων και πόρων για το καταπιστευματικό ταμείο. Προσπαθούμε να συλλέξουμε περισσότερα χρήματα γιατί είναι σημαντική και η παροχή βοήθειας και η παράσταση εκτός από την αποζημίωση. About it, the... δεν έχει δοθεί πολύ μεγάλη δημοσιότητα σε όλα τα θέματα. Για τις Φιλιππίνες όντως ε, έχουμε ε, μια τρέχουσα διαδικασία, δεν πρόκειται να τη σχολιάσω. Ε, αυτό εμπίπτει στην εισαγγελία. και δεν θα ε, έμπαινα ποτέ στα χωράφια της εισαγγελίας. Ήθελα να απαντήσω για τη δικαιοδοσία επίσης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο καταστατικό της Ρώμης είναι ότι η δικαιοδοσία του είναι πάρα πολύ ασυνήθιστη. Μίλησα προηγουμένως για την ε, συμμετοχή, ε, μάλλον για το πώς, ενέχονται οι δράστες είναι συμπληρωματικό το δικαστήριο αυτό και υπακούει στην αρχή της συμπληρωματικότητας. Το καταστατικό της Ρώμης δεν είναι κάτι το οποίο συμφωνήθηκε και είναι στο κενό. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που έχει σχεδιαστεί κυρίως για να ενθαρρύνει τα κράτη είτε μεμονωμένα είτε ως ενότητα κρατών, κοινότητα κρατών, περιφερειακό οργανισμό ή δικαστήρια. Αυτοί φέρουν την κύρια ευθύνη να ε, κάνουν τις ε, ε, έρευνες και να διώξουν τα εγκλήματα αυτά. Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έρχεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει κράτος. Εξού και η καθολική δικαιοδοσία, όπως είδαμε στην υπόθεση της Σενεγάλης. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κράτος ή το κράτος δεν μπορεί να κάνει την έρευνα αυτή, επεμβαίνει το δικαστήριο. Και η μεγαλύτερη επιτυχία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα ήταν να μην έχει ούτε μία υπόθεση, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι διώκονται τα εγκλήματα αυτά στις εθνικές δικαιοδοσίες, τα ίδια τα κράτη. Εξού και η κριτική που ακούμε, αλλά το δικαστήριο αυτό δεν είχε ποτέ ως στόχο να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει τις εθνικές δικαιοδοσίες. Είναι συμπληρωματικό προς τα κράτη. Ε, να περάσουμε στον επόμενο μιλητή αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την ερώτηση για το Συμβουλίο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω αυτό το οποίο συνέβη στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Όταν παραπέμφθηκε η υπόθεση του Σουδάν στο δικαστήριο, το Συμβούλιο ε, είχε την εξή κατάσταση, απήχαν αρκετές μεγάλες δυνάμεις. Αυτό το 2005. Όταν παρέπεψαν την ιστορία για τη Λιβύη το 2010, ήταν ομόφωνη απόφαση ομόφωνη απόφαση το 2011, αρχές του 2011. Ήταν ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει «Α, ε, τώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας υποστηρίζει το δικαστήριο». Ε, εντελώς το αντίθετο. Δεν νομίζω ότι τα μόνιμα μέλη ε, που το Μέιο του 2014 είχαν ένα σωρό βέτο, υπήρχαν κάποιοι άλλοι που είχαν το βέτο στην τσέπη τους για την πρόταση της Ισπανίας να παραπέμψει με την κατάσταση της Σρι Λάγκα στο δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Ένα κράτο μέλος ε, απείλησε να χρησιμοποιήσει βέτο, δεν πήρε το λόγο τελικά, υπήρχαν κάποιες αντίστοιχε περιπτώσει. Τώρα, να δούμε λίγο γιατί κάποιες ε, υποθέσεις δεν προχώρησαν όπως θα έπρεπε. Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, ενέκρινε το 1973 για τη χρήση βίας, το ψήφισμα 1973 υπήρχε το θέμα της χρήσης βίας ε, στην Λιβύη, υπήρχε το προηγούμενο ψήφισμα το οποίο ζητούσε από το δικαστήριο να δράσει, το οποίο δεν ε, ε, εφαρμόστηκε τελικά από το δικαστήριο, το Συμβούλιο, συγγνώμη, το Συμβούλιο δεν είπε ποτέ στις Λιβικές Αρχές ότι εσείς ως καλή αδερφή πρέπει να συλλάβετε και να παραδώσετε τους υπόπτους ε, στο δικαστήριο της Χάγης και να δεχτείτε τα μέτρα για να ενταχθείτε στο καταστατικό της Ρώμης κλπ. Ε, είχαμε ενδείξει μάλιστα στη Χάγη, όχι στη Νέα Υόρκη, ότι κάποιες χώρες μίλησαν στο δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο είναι ανεξάρτητο, επομένως αγνοεί τις προσπάθειες ε, κρατών μελών να παρισφρήσουν στην ανεξαρτησία τους να μην αναλάβουν τις υποθέσεις να τις πάρουν από τη Λιβική δικαιοδοσία. Υπήρχε υπόθεση Ελσενούση, για παράδειγμα, όπου το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Λιβικό Δικαστήριο ε, προέχει. Στην υπόθεση του συνταγματάρχη Καντάφη και τις ε, βίαιες δολοφονίες του Αόπλου ε, ήταν ουσιαστικά εκτέλεση. Είχαμε σαφή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν όχι και έγκλημα πολέμου. Οι μεγάλες δυνάμεις που παρεμβαίνουν στη Λιβύη δεν ζήτησαν από τους Λιβύους να συλλάβουν τον Καντάφη και να τον στείλουν στο δικαστήριο. Δεν θυμάμαι τέτοια δημόσια δήλωση. Υπάρχει λοιπόν πολύ σοβαρό πρόβλημα στο δικαστήριο στο Συμβούλιο, συγγνώμη. Πέραν του γεγονότος ότι υπάρχει συμφωνία τιμωρησίας όπως την αποκαλώ με όσους διαπράττουν ε, πολύ σοβαρά εγκλήματα ε, αποτυγχάνει και το ίδιο το δικαστήριο να δώσει συνέχεια σε αποφάσεις που έχει λάβει το ίδιο για να επεκτείνει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάθεση να αναλάβει δράση το Συμβούλιο. Κατόπιν πρόταση του Λίχτενστάιν και της Μάλτας και άλλων χωρών, από ό,τι φαίνεται, η Γενική Συνέλευση δημιούργησε ένα μηχανισμό για να μπορέσει να διατηρήσει αποδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση της Συρίας που είναι ουσιαστικά μια απελπισμένη κίνηση, αλλά είναι καλύτερη από το τίποτα για να δείξουμε ότι πάνω από 100 χώρες υπερψήφισαν αυτό το ψήφισμα, που σημαίνει ότι μια ψηφοψηφία είναι αυτή η οποία θέλει να διατηρήσει την ατιμορρεσία. Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεσμεύονται για την απόδοση δικαιοσύνης. Ίσως δεν είναι ιστορική στιγμή να συμβεί αυτό εκτός ε, του συστήματος του καταστατικού της Ρώμης, αλλά θα διατηρήσουμε τουλάχιστον τα αποδεικτικά στοιχεία για το μέλλον. Τώρα, το τι θα γίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αυτό επαφίεται σε ε, θεσμούς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια να διατηρήσουν ζωντανή αυτή την κατάσταση ώστε όταν έρθει κατάλληλη στιγμή να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις ανακρίσεις ώστε να τα συγχρηματοδοτήσουν και οι αρμόδιοι διότι το Συμβούλιο είχε πάνω από 100 ψήφους και αυτό είναι πολύ αλλά εάν ζητηθεί από το ε, δικαστήριο να παρέμβει, τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων θα πρέπει να πληρώσουν και όχι οι 100 είναι. Αυτά προβλέπεται από το καταστατικό. Ε, τα επόμενα ψηφίσματα ελπίζουμε ότι θα παραπέμπουν όλες τις περιπτώσεις για οποιοδήποτε έγκλημα. Μπορεί να είναι και τα τέσσερα δηλαδή εγκλήματα και όχι μόνο τα τρία. Ε, μπορεί βέβαια να χρειαστεί να περιμένουμε χρόνια. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και τα κατάλληλα παράθυρα ευκαιρία σε το μεταξύ. Η άλλη ερώτηση ήταν τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να παραπεμφθεί η Ουκρανία στο δικαστήριο. Η Ουκρανία έχει κάνει ήδη αρκετά πράγματα. Έχει αλλάξει το σύνταγμά τη και ε, το έκανε και η Τουρκία η οποία δεν ε, επικύρωσε. Το άρθρο 134 λέει ότι η Ουκρανία μπορεί να αποδεχτεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Το έκανε βέβαια και η Τουρκία πριν από 10 και χρόνια, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί στη συνέχεια. Πέραν αυτού, εφαρμόστη, ε, ε, επιβλήθηκε και μία δέσμη μέτρων, το οποίο δεν συνέταξαν όμως εμπειρογνώμονες για μια μεταβατική διάταξη τριών ετών για να αναβληθεί η εφαρμογή μόνο αυτού του άρθρου μέχρι το 2019 για να προσχωρήσει η Ουκρανία. Δηλαδή όταν δεν θα είναι πια πρόεδρος ο Μποροσέγκα, ίσως να έχουμε κάποιον άλλον, δεν ξέρουμε ποιον. Είναι σαν να δίνουμε την καυτή πατάτα αλλού, στην επόμενη κυβέρνηση. Ε, αυτή είναι πολιτική ποντίου πιλάτου, την οποία δεν θα πρέπει να αποδεχθεί ε, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να, πρέπει να του πούμε ότι πρέπει να άρετε αυτή τη μεταβατική διάταξη. Το δικαστήριο είναι ποινικό δικαστήριο και δεν χρειάζεται να φοβηθείτε τίποτα αν είστε μέλος ε, του δικαστηρίου. Εμείς θέλουμε να προλάβουμε τα εγκλήματα, θέλουμε να σώσουμε τη ζωή θυμάτων και αν το να προσχωρήσει κάποιο στο δικαστήριο μπορεί να σώσει κάποιε ζωέ. Ε, θα πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει λόγος αναβολής. Ο Πρωθυπουργό, για παράδειγμα, του Ιράκ είπε στα μέλη ε, κάποια στιγμή ότι όχι τώρα, αργότερα, γιατί θέλω να λύσω την κατάσταση στη Μοσούλη. Δεν είναι το σωστό επιχείρημα αυτό. Το σωστό επιχείρημα είναι να σώσουμε ζωές όσο μπορούμε και να μην υπάρχει χρήση βίας. Ε, τέτοια δέσμευση θα θέλαμε να δούμε Βεβαίω, ε, ο εκπρόσωπο του δικαστηρίου ξέρουμε ότι έκανε πολύ σημαντική δουλειά, είπα ότι εκπρόσωπο, συγγνώμη, έκανε πολύ σημαντική δουλειά στι διμερεί επαφές στο Κίεβο και γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά ε, συμμετοχή και πολιτικών ηγετών και υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και τις σχέσεις με το Ουκρανικό Κοινοβούλιο που έχετε να τις χρησιμοποιήσετε και γι' αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ας αναφερθώ λοιπόν σε κάποιες από τις εξωτε... εξαιρετικές ερωτήσεις σας. Η κυρία Μπίλερ με ρώτησε αν είχα να δώσω συμβουλές για να πιεστούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν προχωρήσει στην επικύρωση των τροπολογιών της Καμπάλα. Έχουν δει το εγχειρίδιο αυτό και στο εγχειρίδιο υπάρχουν λόγοι για τους οποίους πρέπει κανείς να επικυρώσει. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω στην παρούσα φάση οι βασικοί δισταγμοί έχουν σχέση με την συζήτηση στην οποία αναφερθήκατε πριν, μια τεχνική συζήτηση για τον μηχανισμό opt-out και τι σημαίνει. Θα προσπαθούσα να το θέσω αυτό όχι με τεχνικό τρόπο. Κάποιες χώρες ανησυχούν σχετικά με το ποια είναι η νομική τους κατάσταση σε σχέση με μια χώρα η οποία δεν έχει επικυρώσει την τροπολογία. Η απάντηση σε αυτό είναι σαφής. Αν επικυρώσεις την τροπολογία, δεν έχεις πια αυτή την ανησυχία. Είναι σαφές λοιπόν αυτό και ισχύει το ότι ορισμένες χώρες που έχουν επικυρώσει τις ε, τροπολογίες, έχουν κάνει και συζητήσεις για το τι σημαίνουν οι τροπολογίες αυτές, λέγουν ταυτόχρονα ότι δεν θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις τώρα, γιατί έτσι και αλλιώ αφορά κράτη τα οποία δεν έχουν επικυρώσει. Είναι ένα επιπλέον επιχείρημα δηλαδή και ίσως κάπως πιο σοβαρά να πούμε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Είμαι βέβαιος ότι θα ολοκληρωθούν στο τέλος του χρόνου και στη συνέχεια θα υπάρξουν κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις χώρες αυτές να ολοκληρώσουν την διαδικασία σε εσωτερικό επίπεδο. Εγώ όταν είπα εύκολο να προσαχθούν ή μάλλον εύκολο να ξεκινήσει η διαδικασία η δικαστικής βάρος τους, αυτό το οποίο εννοώ δεν ήταν σωστό βέβαια, είναι ότι ίσως να μην είναι και τόσο πολύ δύσκολο να διωχθούν οι χώρες αυτές, γιατί ο ορισμός της επίθεσης στοχεύει ακριβώς σε αυτό το οποίο κάνει ο ηγέτης μιας πλευράς και δεν πρέπει να χρειαστεί να πάει κανείς στο πεδίο μάχης ή επιτόπου και να συλλέξει στοιχεία για το τι εγκλήματα έχουν γίνει και μετά να διατυπώσει την καταγγελία, την δίωξη είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να μάθει ακόμα και από τη δημόσια ρητορική των συγκεκριμένων ηγετών που σαν παραδείγμα ζητούν και προκαλούν την παράνομη χρήση βίας. Όταν αναφερθήκατε στη Νιρεμβέργη φυσικά δεν ήταν εύκολα τα πράγματα εκεί. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα εδώ για την δίωξη των πλευρών. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε πάντα την υπόθεση από πλευράς ε, των, ε, της υπεράσπισης και όσο χαμηλότερα κατεβαίνει κανείς στην αλυσίδα αν θέλετε της εξουσίας, τόσο πιο δύσκολο είναι να αποδείξει κανείς ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι υπεύθυνο για μια πράξη επίθεσης. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με έναν ηγέτη, τότε μπορούμε τη δίωξη να την ασκήσουμε με κάπως ευκολότερο τρόπο. Οπότε είναι δικαιολογημένη τώρα η χρήση βίας και πότε όχι. Να τονίσω εδώ από τη μία ότι στα πλαίσια του ορισμού ακριβώς της επίθεσης η χρήση βίας για λόγους άμυνας και που τεκμηριώνεται από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μία επίθεση και να διωχθεί. Ε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες ρήτρε που λέγουν ότι μόνο οι πιο ξεκάθαρες μορφές επίθεσης είναι ε, οι πιο προφανείς, αυτές θα πρέπει να διώκονται από το Διεθνές Δικαστήριο με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο σαν κατηγορούμενο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιες άλλες πλευρές, κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες δράσεις δεν είναι παράνομες. Αλλά το να παραπέμψουμε τον ηγέτη μιας χώρας στο δικαστήριο γιατί έχει διαπράξει το έγκλημα του, της επίθεσης είναι το μέγιστο δυνατό μέσο το οποίο έχουμε στην διάθεσή μας και από την άλλη είναι κάτι το οποίο μας επιτρέπει να συμφωνήσουμε στον ορισμό της πράξης. Το θέμα δεν είναι να συμμετέχουν στην απόφαση αυτή μόνο τα μέλη του δικαστηρίου, αλλά και μια ομάδα εργασίας στην οποία να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Και όταν έγινε δεκτή η πρόταση, όλα τα κράτη-μέλη συμμετείχαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι ήταν εύκολο μόνο το κομμάτι των ανώτατων στελεχών στην Χαϊδελβέργη. Τώρα δεύτερος γύρος. Δεν ξέρω αν κάποιο θέλει το λόγο. Κυρία Γκόμε, ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι την υπηρεσία εξωτερική δράση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν μπορούν να μα πούν τι κάνουν για να υποστηρίξουν την κοινωνία των πολιτών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της ατιμορρησίας για να προσάγονται στη διεθνή δικαιοσύνη, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι ένοχοι, οι όταν ε, στη Συρία έχουμε προφανείς παραβιάσεις ε, ε, και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Και πώς υποστηρίζουμε κάποιους που συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία επιτόπου για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα και να φτάσει στη δικαιοσύνη. Όπως γίνεται με τους Γεζιντή που ήταν θύματα γενοκτονίας. Νομίζω ότι εσείς μπορείτε να παίξετε πρωταγωνιστικό ρόλο υποστηρίζοντας έμεσα και άμεσα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τους φορείς επιτόπου, για να μην μιλήσω για την πολιτική υποστήριξη με τις αρχές διαφόρων κρατών, όπως ήδη ακούσαμε από τον κύριο Ντόνατ Κάτιν. Και επίση θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς το βλέπει το δικαστήριο έχει κανένα ρόλο συμβουλευτικό ή άλλο στη δίκη του Ισένα Μπρέ στη Σενεγάλη που μόλις επιβεβαιώθηκε από ένα φετίο. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό, η αλλο στη δικη του ισενα μπρεστη στη σενεγαλη που μολις επιβεβαιωθηκε απο ενα φετιο ηταν πολυ σημαντικο αυτο η καταπολεμηση της ατιμορρησίας, όπου ένα κράτος μέλος αποφάσισε να θέσει στην υπηρεσία σας το ε, δικαστικό του σύστημα. Υπήρχε συνεργασία ε, σε αυτό το τομέα και σε άλλες δίκες. Πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις. Μήπω με την αντίστροφη σειρά, αν έχετε να σχολιάσετε κάτι, ο κύριος Μπαρίγκα, όχι. Περισσότερες μάλλον είναι για την κυρία Πρόστ. Για το τελευταίο. Για τη δίκη αυτή στη Σενεγάλη. Είναι πραγματικά ένα εύγλωτο παράδειγμα για το πώς εφαρμόζεται το καταστατικό της Ρώμης. Με την, εκτεταμένη, την επέκταση μάλλον της δικαιοδοσίας, ένα κράτος ανέλαβε την ευθύνη να ε, προχωρήσει στην ε, συγκεκριμένη δίκη. Εδώ μπαίνει η αρχή της συμπληρωματικότητα. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο υποστήριξε όλη αυτή τη δίκη και τουλάχιστον δύο ή τρεις δικαστές ήταν παρόντες ε, στην ε, αρχή της δίκης για να δείξουν ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα του καταστατικού της Ρώμης. Δεν είμαι βέβαια αν υπήρχε ε, συγκεκριμένη συνεργασία ουσιαστική αλλά έχουμε επανειλημμένα περιπτώσεις όπου γίνονται έρευνες και διώκεται ένα έγκλημα και τοπικά αλλά και σε συνεργασία με το δικαστήριο όπως συνεργαζόμαστε με τις εθνικές δικαιοδοσίες, στις έρευνες και στη δίωξη των εγκλημάτων αυτών. Είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτό και πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει σχεδιαστεί το όλο σύστημα του καταστατικού της Ρώμης. Κύριε ε, Ντονάτ Κάτσεν, ναι, θέλω να επανέλθω σε ένα μόνο σημείο που αναφέρθηκε για το θέμα της Αφρικής και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα ήθελα να τονίσω ότι το κύμα αποσύσεων που είδαμε πέρσι τον Οκτώβριο προκάλεσε τέτοια σφοδρή αντίδραση από την κοινωνία των πολιτών, εθνική και διεθνή, και σε συνεργασία με ΜΚΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους, καταφέραμε πραγματικά να αναστρέψουμε αυτή την ε, πορεία. Θα ήθελα εδώ να σχολιάσω με περηφάνεια το γεγονός ότι το Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή της Νότιας Αφρικής ε, ζήτησε ε, να ανατραπεί η κατάσταση. Είχε ζητήσει η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ε, να καταργηθεί η νομοθεσία με ένα νέο νομοσχέδιο και με την πρωτοβουλία του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου κατάφεραν να αποσυρθεί αυτό από το Κοινοβούλιο και είπαν ότι ε, ε, Δία πάντως έχει αυτό διαγραφεί από την κοινοβουλευτική μας ε, πρακτική. Δεν θέλουμε να έχουμε πιστοδρόμηση. Υπήρχε το Ε, το, αντίστοιχο κέντρο ε, στην Νότια Αφρική είπε ότι το γεγονός ότι δεν κατάφερε να συλληφθεί το 2015 ο πρόεδρος Μπασίρ του Σουδάν ε, οφεί, οφείλεται αυτό ότι ήταν ε, αντίθετο με την ε, νομοθεσία της Νότιας Αφρικής. Στην Κάμπια αντίστοιχα είδαμε και τώρα συνεργαζόμαστε με τους βουλευτές της χώρας για να μην έχουμε φαινόμενα τύπου Νότιας Αφρικής ε, να επαναλαμβάνονται. Μπορεί η κατάσταση να είναι περίπλοκη, αλλά ήθελα να, πω, για, να ακουστεί και να σημειώσετε. Έχει ανατραπεί αυτή η πορεία που είχαμε διαπιστώσει το πέρσι το φθινόπωρο. Και για να τελειώσω, την περασμένη εβδομάδα η Βουλή του Νίγηρα προσκάλεσε την εισαγγελέα μας, την εισαγγελέα μάλλον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και αποκατέστησε τη ε, σχέση της με την κοινωνία των πολιτών ε, έκανε έντονη την παρουσία της. Αυτά όλα είναι μια ε, προσπάθεια πάγια και διαρκής, γιατί τελικά το μήνυμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κερδίζει έδαφος, πείθει την κοινή γνώμη και στην Αφρική και αλλού και εκείνοι που θέλουν να μποϊκοτάρουν το έργο και να το συσκοτήσουν και να το αμαυρώσουν δεν επιτυχάνουν στην προσπάθεια αυτή. Fantastic. Ε, Εξαιρετικά. Υπήρξε και μία εν μέρη ερώτηση προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θέλετε το λόγο. Ωραία. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει με πρακτικό επιχειρησιακό τρόπο το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Υπάρχει ισχυρή δέσμευση και απόφαση του Συμβουλίου του 2011 και πρόγραμμα δράσης, δηλαδή εξηγούνται τα πάντα ό,τι κάνουμε για το δικαστήριο. Και όσον αφορά τη χρηματοδότηση, Έχουμε περίπου 37 εκατομμύρια ευρώ από το 2000 ε, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί είτε για άμεση στήριξη του δικαστηρίου ή για την κοινωνία των πολιτών η οποία υποστηρίζει το καταστατικό της Ρώμης. Ε, μόλις υπεγράφηκε μια νέα σύμβαση όπως γίνεται κάθε χρόνο με το δικαστήριο για να συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη για το 2016 και το 2017. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν προωθεί και αυτή το καταστατικό της Ρώμης ε, μέσω άμεσης χρηματοδότησης του δικαστηρίου. Επίσης ε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτοί που αξιολογούν το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που είναι η βασική ε, πηγή στήριξη. Μόλι εξέδεσαν μια έκθεση, πρόκειται για ανεξάρτητη αξιολόγηση βεβαίω, η οποία επισημαίνει και αυτή τη σημασία να συνεχιστεί η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της ατιμορρησίας και του δικαστηρίου βεβαίως, που σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η υποστήριξη ε, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το μέσο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή ακρόαση για το θέμα αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις πολύ για τον χρόνο σας. Πρόκειτο για μια ενημέρωση υψηλού επίπεδου και σας ευχαριστώ που βρήκατε το χρόνο και κάνατε και τον κόπο να έρθετε εδώ στην Επιτροπή μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερη προσέλευση βεβαίως, αλλά αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε στο μέλλον, να δούμε ποια είναι η κατάλληλη σύνθεση για να το κάνουμε αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν ε, ε, αντανακλά ε, το ενδιαφέρον που έχουμε στην πραγματικότητα για την παρουσίαση εδώ και τα όσα είχατε να μας πει. Με αυτά ολοκληρώσαμε για σήμερα. Αύριο έχουμε συνεδρίαση διευρυμένου Προεδρείου στις 9 και η Επιτροπή θα συνεχίσει στις 10. Πέρα συνεδρία. Σας ευχαριστώ για σήμερα.